στην συνεδρίαση. Πρώτα, να εξετάσουμε τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίασης. της 22ης δηλαδή Οκτωβρίου 2009. Ε, αν τα εγκρίνετε, εγκρίνονται λοιπόν αφού δεν είσατε κανείς. Προχωρώ στο τρίτο θέμα της σημερινής διάταξης που θα είναι και πιο σύντομο από ό,τι την προηγούμενη φορά. Θα σας πω λίγα ενημερωτικά για θέματα τα οποία, για γεγονότα τα οποία ε, συνέβησαν μετά από την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι σήμερα. Το γραφείο Ζαχάροφ που θα απονεμηθεί στις 16 ε, Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Έχω μια πρόσκληση να μεταβώ στην Μόσχα σε μια διάσκεψη πριν από αυτή την ημερομηνία το Ίδρυμα Ζαχάροφ οργανώνει διάσκεψη για την κληρονομιά του βραβείου Ζαχάροφ και είναι η επέτειος ε, του θανάτου του ε, Ζαχάροφ θα μπορέσουμε να ε, συναντηθούμε και με τους φίλους μας στο Στρασβούργο μετά από τη διάσκεψη της Μόσχας. Θα σας τηρώ ενήμερους πάντοτε, πάντως την προηγουμένη Δευτέρα συναντήθηκα με τους πρέσβεις των 27 χώρων μελών και ο Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ πρόεδρος της Επιτροπής Λίμπε ήταν επίσης παρόν και γνωρίζετε ότι η δική τους, ο δικός τους κύκλος αρμοδιοτήτων έχει σχέση με τα εσωτερικά ε, ανθρώπινα δικαιώματα, την περιθωριοποίηση κλπ. Ενώ στη δική μας υποεπιτροπή ασχολούμαστε περισσότερο με την εξωτερική πτυχή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η συζήτηση με τους πρέσβεις που εκπροσωπούν το, εκπροσωπούσαν την προκειμένου το Συμβούλιο των Υπουργών ήταν καλή. Ζήτησαν οι πρέσβεις να μάθουν τη δική μας άποψη σε σχέση με την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό θα μας απασχολήσει πολύ όλο το χειμώνα στην Υποεπιτροπή μας. Ο στόχος δεν είναι η Επιτροπή Συνταγματικών να συντάξει μια γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας σχετικά με την προσχώρηση της Ένωσης στην Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εμείς θα έχουμε βεβαίως κάποιο ρόλο να παίξουμε στην διαδικασία αυτή. Μπόρεσα λοιπόν τουλάχιστον να κάνω μια δήλωση σχετικά με αυτό το θέμα. Και βέβαια η συνθήκη της Λισαβόνας αρχίζει να εφαρμόζεται από αύριο. Επομένως και αυτή θα έχει ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο και θα μας επιτρέψει επίσης να προσχωρήσουμε στην Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαι βεβαίω ότι τα εγγόνια μας δεν θα μας ρωτήσουν απαραίτητα πότε ε, ε τέθηκε σε ισχύ ή αξιονεφαρμόζεται η συνεφαρμόζεται η συνθήκη της ε, Λισαβόνας και που ήμασταν εκείνη την ώρα. Τώρα η Βαρόνη Άστον που είναι η νέα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και θα είναι η πάτη εκπρόσωπος. Ε, αυτό εμένα με ικανοποιεί πολύ. Ε, γνωρίζω ότι ενδιαφέρεται πολύ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί της την Τετάρτη το πρωί που θα προσέλθει στην Επιτροπή Εξωτερικών για ανταλλαγή απόψεων θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε ποια είναι η γνώμη της για το mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ένταξή τους δηλαδή ως πτυχή σε όλα τα θέματα. Και τώρα για τα κατεπήγοντα, την προηγουμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε Νικαράγουα, Λάος και Βιετνάμ και Κίνα. Είχαμε αυτά τα επίγοντα ψηφίσματα. Ίσως σημειώσατε ότι το Κοινοβούλιο δεν συμφωνεί απαραίτητα. Δεν είναι δηλαδή όλα τα μέλη του σύμφωνα με τη στάση μας, με, μια ενιαία στάση απέναντι στην Κίνα ή στην Ικαράγουα. Θα συζητήσουμε λοιπόν ξανά μέχρι ότου εναρμονιστεί η ε, στάση μας. Σχετικά με αυτά τα ψηφίσματα της Πέμπτης το απόγευμα, Και σε αυτά θα έχει αντικτύπω η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα γίνουν δηλώσεις σχετικά και νομίζω, ελπίζω μάλλον, ότι θα γίνουν αυτές και σε υψηλό επίπεδο. Και θα σας θυμίσω ότι έχω αποστείλει επιστολή στους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων ήδη από τα τέλη του καλοκαιριού και ίσως θα καταστεί δυνατόν να προωθηθεί η, η συζήτηση αυτή. Ο κύριος Ομπιόλς είναι παρόν και θα μπορέσει να εξηγήσει λίγο ε, το ταξίδι που έκαναν στην Μαδρέτη στα τέλη Οκτωβρίου με την αντιπροσωπεία. Η Ισπανία λαμβάνει τώρα την Προεδρία και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τη ε, σημασία αποδίδει στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την περίοδο της θητείας της. Θα ακούσουμε και από τον κ. Χάουιτ ή ίσως από την κυρία Αντρικιένε που συμμετέσχουν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προ λίγων εβδομάδων. Και το θέμα αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε εκεί που θα συζητήσουμε μετά της Σουηδικής Προεδρίας. Εξαρτάται από τη γνώμη που έχουν οι ε, κύριοι Χάουιτ και Αντρικιένε. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο υπαριθμό 4 που προβλέπει ανταλλαγή απόψε με τη Σουηδική Προεδρία. Νομίζω ότι μείναμε όλοι ικανοποιημένοι και εγώ ε, Χάρηκα πολύ τη συνεργασία με την Σουηδική Προεδρία, η οποία έχει σαφέστατη γνώση των θεμάτων των θεπιών δικαιωμάτων και η κυρία Σάμερ Σιόλτ που είναι ε, πρόεδρος της ΚΟΧΟΜ ήταν σε στενή συνεργασία πάντοτε με την υποεπιτροπή μας. Τώρα, η Ισπανική Προεδρία που θα αναλάβει την ΚΟΧΟΜ δηλαδή, ο, ο, ο πρόεδρος της θα είναι ο κύριος Φερνάντο Ερέιρα που είναι της μόνιμης ισπανικής, ερέδια, που είναι της μόνιμης ισπανικής ε, ε, αντιπροσωπείας και θα αναλάβει. Δυστυχώς ε, η ίδια η Ισπανική Προεδρία δεν μπορεί να είναι παρούσα, αλλά ο κ. Φερνάντο Ερέδια είναι παρόν. Η νέα Προεδρία της ΚΟΧΟΜ έχει προσκληθεί να προσέλθει στις 14 Ιανουαρίου στην συνεδρίαση της υποεπιτροπής μας. Θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τότε την ε, συζήτηση και με την Ισπανική ε, Προεδρία. Έχουμε και την Νατάλια Αλόνσο παρούσα, η οποία εκπροσωπεί την Διεθνή Αμνηστία, το Γραφείο Βρυξελών. Κατά τις αρχές της Σουηδικής Προεδρίας εξετάσαμε το φιλόδοξο πρόγραμμά τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Σουηδοί επιζητούσαν μια πιο συνολική προσέγγιση ε, για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλές από τις κατευθυντήριες γραμμές και τον διάλογο και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Σουηδία για την υποστήριξη της δημοκρατίας και για να καταστεί πλέον ορατή η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην παρουσίαση του φιλοδόξου προγραμματός της η Σουηδική Προεδρία είχε δηλώσει τότε ότι επιθυμούσε να γίνει πλέον αποτελεσματική χρήση των υφισταμένων μηχανισμών, να γίνει και το λεγόμενο mainstreaming σε όλο το φάσμα δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα παρακαλέσω την κυρία Χάμαρ να λάβει το λόγο και να μας εξηγήσει πώς εφαρμόστηκε το πρόγραμμα αυτό στη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας και θα ακούσουμε επίσης και για το ψήφισμα. που έγινε ε, δεκτό, που εγκρίθηκε δηλαδή στο Συμβούλιο στις 16-17 Νοεμβρίου. Κυρία Χάμαρσκιολτ και πάλι με χαρά σας βλέπουμε κοντά μας και σας δίνω μέσω τον λόγο. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που βρίσκομαι πάλι εδώ. Καλά θα ήταν να αλλάξει μικρόφωνο για κυρία Χαμάρσκιολτ, γιατί είναι λίγο μακριά αυτό που έχει ανοιχτό τώρα. Η... Ίσως είναι συμβολικό το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας στις 30 Νοεμβρίου. Και όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, ε, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αύριο η συνθήκη της Λισαβόνας και θα μας εισαχάγει έτσι σε ένα νέο κεφάλαιο της, Ευρωπαϊκής, της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα πάντως θέλω να σας εξηγήσω τα πράγματα που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο μας. Μένει ακόμα να κάνουμε πολλά. Είμαι στη διάθεσή σας βέβαια να ε, να συζητήσω μαζί σας μαζί και με τους συναδέλφους μου της Προεδρίας και του Συμβουλίου. Η στρατηγική της Σουηδικής Προεδρίας στον τομέα αυτό ήταν προορατική και αυτό δείχνει επίσης ότι αυξάνεται συνεχώς το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Από την εμπειρία μα από τους προηγούμενους μήνες ε, βλέπουμε ότι ο αυξανόμενος ρόλο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασίζεται στι κοινέ προσπάθειε ε, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι είχαν κρίσιμη σημασία για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Του τελευταίους μήνες το Συμβούλιο είχε διάφορες ευκαιρίε σε διάφορα επίπεδα για να κάνει ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα με την Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία. Χαίρομαι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε, επίσημα και εμεί, δημόσια και εμπιστευτικά, που έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν και συνεισφέρουν στις προσπάθειες που κάνουμε, ούτω ώστε ο ρόλο Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο ορατό και πιο συνεκτικός στο μέτρο τη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων. Τους τελευταίους μήνες έχουμε εστιάσει την προσοχή μας σε διάφορα ζητήματα που κρίνουμε σημαντικά και εμείς και το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, ε, ως Προεδρία εστιάσαμε την προσοχή μας στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο τοπικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αντιδράσει. Όταν διαπιστώσαμε συγκεκριμένες παραβιώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε διατηρήσει επαφέ με του επερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με άλλου μη κυβερνητικέ οργανισμού σχετικά με τι βέλτιστες στρατηγικέ που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε ε, πολύ σημαντικέ ε, περιπτώσει. Ε, βέβαια υπολείπεται μεγάλο έργο. Επίσης, στη Ρώσια οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απομονήμει στο Memorial και σε άλλου υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το βραβείο Ζαχάροφ. Επίση έχουμε δράσει στο Ιράν, στην Κίνα, στο Ιράκ, στην στην Κολομβία, στο Καζανκστάν, στη Σιμπάμπουε, στη Σρι Λάγκα και στην Κούβα σε συνεργασία με τους εκεί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ως Προεδρία εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειες που κάνουμε για τις επικαιροποιημένες κατευθυντηρίες γραμμές ε, για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατάσταση των ομοφιλοφίλων, αμφιλοφίλων και τρανσέντερ Ε, κυρίως σε σχέση με την ε, χρήση πληροφοριών στο ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, υποστήριξη της δημοκρατίας. Στις 17 Νοεμβρίου ενέκρινε το Συμβούλιο συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας και σε σχέση με την ΚΕΠΑ και σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά τα συμπεράσματα ενέχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα σχετικά με την ιεράξη των προτεραιοτήτων και τη συνοχή της πολιτικής μας. Ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα και ε, η ατζέντα δράσης θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία, εργαλεία που έχει στη διάθεσή τη ε, για να εφαρμόσει μια συνεκτική στρατηγική. Επίση, έχουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 22η Οκτωβρίου σχετικά με αυτέ τι προσπάθειε, όπου τονίζεται η σημαντική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώ και των εθνικών και περιφερειακών βουλών ε, ω προ την υποστήριξη τη ε, προσπάθεια του εκδημοκρατισμού. Τρίτον, θα θέλαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στι ειδικέ ανάγκε πριν από λίγες ημέρες, στις 26 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε το συμπέρασμα της Ευρωπαϊκής ε, Κοινότητας ε, σχετικά με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Ε, όλοι περίμεναν εδώ και καιρό αυτή την κίνηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι η πρώτη φορά που μια περιφερειακή οργάνωση προσχωρεί στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα άλλο θέμα τώρα, η σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις. 10 και 11 Νοεμβρίου συγκάλεσε η Σουηδική Προεδρία μια συνεδρίαση με τίτλο «Προστασία τήρηση των δικαιωμάτων και ένδικα μέσα», δηλαδή μια διάσκεψη σχετικά με την κοινωνική εταιρική ευθύνη, ε, όπου παρευρέθηκε ο ειδικό ηγετής του ΟΗΕ, ο κ. Τζον Ράτζι. Κύριε Πρόεδρε, ε, ένα γενικό στόχο τη Σουηδική Προεδρία ήταν να διατηρηθεί η θέση που κατέχει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ω βασικό παγκόσμιο παίκτη στον τομέα αυτό. Θέλουμε να προάγουμε, να καταστήσουμε πιο εμφανείς τις στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηλώνουμε ικανοποιημένοι διότι η Πολιτική Επιτροπή και η Επιτροπή ασφαλεία το Σεπτέμβριο ενέκρινε μια σειρά μέτρων ε, για να προάγει το ρόλο και την εικόνα τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τη βάση εξαιρετικών προτάσεων που έκανε η Γραμματεία του Συμβουλίου Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα παραδείγματα, αυξημένη χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πιο συστηματική δημοσίευση των δηλώσεων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα φόρα και επίσης καλύτερη κάλυψη της μεμονωμένης κατάσταση αναχώρα δηλαδή, καθώς και την ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν από το τέλος της Σουηδικής Προεδρίας θα έχουμε περατώσει 17 διαλόγους και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό την αιγίδα της ΚΟΧΟΜ με χώρες όπως Ρωσία, Κίνα, Καναδά, Καναδά, η Ιαπωνία, η ΙΠΑ, Γεωργία, Κυργιστάν, Τατζικιστάν, Καζακστάν, Αργεντινή, Βραζιλή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Μεξικό, με τις υποψήφιες χώρες και με την Αφρικανική Ένωση. Χαιρόμαστε που θα διοργανώσουμε την πρώτη συνεδρίαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αρμενία στην ιστορία στις 8 και 9 Δεκεμβρίου και να αναφέρω επίσης ότι τον Οκτώβριο αποφάσισε το Συμβουλίο να δρομολογήσει νέο διάλογο με την Ινδονησία. Δρομολογήθηκε ο διάλογος τον Νοέμβριο από τους ε, υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας και της Ινδονησίας. Πέραν αυτού, σε πολιτικό επίπεδο θέτει διαρκώς το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Συμβούλιο και ε, μεταξύ άλλων και στην έσχατη σύνοδο ε, ε, ε, με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο διάλογος αυτός και οι διαβουλεύσεις είναι στοιχείο κλειδί της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο απότερος στόχος είναι να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Σε αυτά τα πλαίσια αρχίσαμε την αξιολόγηση του διαλόγου ΕΕ Κίνα που, στην οποία προαναφέρθηκα και θα ενημερώνουμε διαρκώς την Οικοεπιτροπή για την πρόοδο που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Πέρα από το διάλογο και τις διαβουλεύσεις που διοργανώνει η όπως έχουν διοργανωθεί διάφορες άλλες ε, συνεδριάσεις ε, για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε άλλα φορά, επί τη βάση παραδείγματος χάρη του άρθρου 8 της Συμφωνίας του Κότονου. Παραδείγματος χάρη η Συμφωνία με τη Ζιμπάμπουε για να συνεχιστεί ο διάλογος του άρθρου 8 ε, και άλλες συνεδριάσεις ε, με τους νότιους γειτονές μας, ε, με την Παλαιστινιακή Αρχή, με το Ισραήλ, με το Μαρόκο και με την Αίγυπτο, στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. τώρα, Σχετικά με, ε, πιστεύουμε ότι η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ε, έχει ως αποτέλεσμα να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Από την αρχή της Προεδρίας μας έχουμε κάνει διάφορες παρεμβάσεις σε πάρα πολλές χώρες άνω τον κόσμο και έχουμε κάνει περίπου 12 διαβήματα και σχετικές δηλώσεις για την κατάσταση στις συγκεκριμένες χώρες. Σε σχέση με την θανατική ποινή, η Προεδρία μας συνέχισε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργησή της, ε, αντιδρώντας σε εκτελέσεις που είχαν ε, προβλεφθεί σε διάφορες χώρες. Γιορτάσαμε την Ευρωπαϊκή μέρα κατά της θανατικής ποινής 10 Οκτωβρίου μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, και τονίσαμε και στη Γυναική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτό το θέμα σε μια δημιουργική συνάντηση και επίσης σε δύο εβδομάδες θα γιορτάσουμε τη 15η επέτειο του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασή. Για τα βασανιστήρια αντιδρούμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις και συνεχίσουμε να προάγουμε την επικύρωση του ε, προαιρετικού πρωτοκόλλου της σχετικής σύμβασης του ΟΗΕ για την κατάργηση των βασανιστήριων. Εντατικοποιούμε τις διμερείς δράσεις μας βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών ε, και βάσει των συστάσεων ε, των συμβαλωμένων μερών του ΟΗΕ. Όπω γνωρίζετε, έχουμε δρομολογήσει δράση για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ε, στο Φόρουμ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στι συνεδρίε που διοργανώθηκε στο Χόλμη σε 6 και 7 Ιουλίου για την, για την καταπολέμηση τη βία κατά των παιδιών. Έχει εκδοθεί πλέον και η ε, τελική έκθεση από αυτή τη συνεδρία και είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του Φόρουμ. Επίση, η ΚΟΧΟΜ το Δεκέμβριο θα συναντηθεί με την κυρία Μάρτα Σάντο δηλαδή την ειδική εντεταλμένη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Τώρα για τις κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα των παιδιών και για τις ένοπλες σειράξεις, το Συμβούλιο έχει εντοπίσει συγκεκριμένες χώρες και πιλωτικές δράσεις ε, προς τα... και θα κατευθύνουμε τη δράση μας ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε αναλάβει διάφορες ε, δράσεις, παραδείγματο χάρη μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την εφαρμογή σχετικής σύμβασης στο Χόλμη τον Νοέμβριο και σε τοπικό επίπεδο έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες σε τρίτες χώρες χώρες ε, μέσω των πρεσβειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρυσι εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές επίσης για τη βία και την διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών και των κοριτσιών και το καθήκον της, Ευρωπαϊκής, της Σουηδικής Προεδρίας ήταν να καταστήσει λειτουργικές αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές. Προς το παρόν έχουμε πάρει από τους επικεφαλείς των απόστολων μας εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή αυτών των κατευθυντριών γραμμών από πάνω από 80 χώρες και τώρα ε, επεξεργαζόμαστε ε, ε, τις εκθέσεις αυτές για να καταλήξουμε καταλήξουμε σε συμπεράσματα ε, και επίσης η επέτειος ε, της σύμβαση DAW μας δίνει μια ευκαιρία να θίξουμε το θέμα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα των γυναικών. Διάλογο που έχουμε με τρίτες χώρες και με την Αφρικανική Ένωση μεταξύ άλλων επίσης. Ενισχύουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εργασίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορες διεθνούς οργανισμούς, διεθνούς οργανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συντονίζουμε διαβήματα σε διάφορες χώρες, ε, ε, κυρίως ε, όπου έχουν σημειωθεί ένοπλες σειράξεις, επί τη βάση των κατευθυντήριων γραμμών IHL επίσης. Έχουμε την 60η επέτεια των συμβάσεων της Γενέβης και οργανώσαμε σε Βρυξέλλου Σεπτέμβριο μία διάσκεψη για τον εορτασμό της επέτειου για να συνεχίσουμε την προαγωγή των θέσεων της ευρωπαϊκή Ένωσης ε, σε σχέση με την ICC. Τα τελευταία χρόνια επίσης ε, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος ε, για την ενσωμάτωση στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου. Και ε, θέλουμε να υπάρχει συνοχή στι ε, πολυμερεί προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με, χάρη, με τον ΟΑΣΑ, με τον ΟΗΕ, με το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Στην ιστοσελίδα μα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των ε, διαβουλεύσεων. Επίση, ζητήσαμε από τον εκπρόσωπο Κιόνκα να ε, μεταβεί στο Στρασβούργο και στην Βιέννη, ώστε να δούμε στα πλαίσια αυτών ε, των βημάτων πώς μπορούμε να προάγουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και σχετικά με την ΚΕΠΑ θέλουμε να ενσωματώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και την ανάλυση προκύπτει από το AHL στην διοργάνωση των αποστολών μας και στην, για να προάγουμε τη συνειδητοποίηση της κατάσταση σε κάθε χώρα, όπω παραδείγματο χάρη στην Γεωργία. Τον Οκτώβριο τα κράτη-μέλη και κάποιοι προσκεκλημένοι έκαναν την πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του ψηφίσματο του ΟΗΕ 1325. Τώρα, για τα ε, συντηρητικά μέτρα, ε, ε, στιάσαμε την προσοχή μας στο Ουσμπεκιστάν. Δεν αποφασίσαμε να παρατείνουμε τον Οκτώβριο αυτά τα μέτρα, αλλά παρόλα αυτά το Συμβούλιο θέλει να διατικοποιήσει τον διάλογο με, τον με το Ουσμπεκιστάν, κυρίως ε, επιθεωρώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. και μην ξεχνάμε και την αναθεώρηση της διαδικασίας για τις γενικές προτιμήσεις σε σχέση με την Σρι Λάνκα. Ας περάσουμε με τώρα στις ε, πολυμερείς προσπάθειες. Ε, προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να προάγουμε το ρόλο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το ρόλο τους βημάτων λοιπόν για να υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μπορούμε να παρέμβουμε σε κρίσιμες περιπτώσεις. Συνεργαζόμαστε βέβαια με άλλους εθνικούς φορείς και πιστεύουμε ότι με αυτή την διεύρυνση των προσπαθειών μας σε όλα τα επίπεδα έχουμε ε, επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επίσης, ε, πριν ε, από λίγες εβδομάδες είχα ενημερώσει την Υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα για αυτή την κατάσταση. Σήμερα θα ήθελα απλά να τονίσω ότι Ε, είναι σημαντικό να πράγουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, και να αντιδρούμε με τον κατάλληλο τρόπο όταν προκύπτουν σοβαρές παρεμβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2011 θα γίνει η αναθεώρηση του ρόλου του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΕ, όπως ξέρετε, και σε στενή διαβούλευση με τις επόμενες προεδρίες έχει αρχίσει και η δική μας προεδρία της με διάφορους εταίρους για αυτή την αναθεώρηση. Τώρα όλες οι τέσσερις, ε, τα τέσσερα ψηφίσματα του ΟΗΕ έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραδείγματος χάρη το ψήφισμα για τα δικαιώματα του παιδιού που, παρουσίασε η που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η ομάδα λατινοαμερικανικών χωρών ε, νεκρήθη με ομοθυμία για πρώτη φορά από το 2001 Επίσης ε, εγκρίναμε και το ψήφισμα για το Ιράν που υπέβαλε ο Καναδάς. Ε, δεν υπήρξαν ε, αντιπροτάσεις κατά των ψηφισμάτων φέτος και θεωρούμε ότι αυτό είναι θετικό. Επίσης δεδομένου του ευρύτερου κλίματος για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ρατσισμού και της θρησκείας έχουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Ένωση για την κατάργηση όλων των μορφών της διακριτικής μεταχείρισης και που εγκρίθηκε με επίσης αριθμό ρεκόρ κόσπων ε, δηλαδή από ε, μεγάλο αριθμό των χωρών, συγκεκριμένα 82. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πάρα πολλά κράτη καταψήφισαν το ψήφισμα του ΟΗΕ σχετικά με την συκοφαντική δράση κατά συγκεκριμένων θρησκειών. Τώρα, Ε, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα όσων έχουν αλλάξει φύλλο ε, συνιστά προτεραιότητα για μας ε, και στις 10 Δεκεμβρίου που είναι η ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θα διοργανώσουμε μια παράλληλη εκδήλωση από πλευράς Προεδρίας ε, και συνεργαζόμαστε με οργανώσεις ε, προστασία των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων για να εντατικοποιήσουμε και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και θα συνεχίσουμε να έχουμε ενεργό ρόλο για την καταπολέμηση του ρατσισμού ε, και κάθε μορφής διακριτικής ε, μεταχείρισης. Ε, δηλώνουμε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των εργασιών της διακυβερνητικής ομάδας για την εφαρμογή της δήλωσης του ντουρμέν και το σχετικό πρόγραμμα δράσης. Παρόλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις στη Γενική Συνέλευση χαρακτηρίζονταν από, ισχυρή πόλωση και αυτό το φθινόπωρο. Όταν μίλησα στην υποεπιτροπή σας τον Αύγουστο, ε, τόνισα ε, ότι η Προεδρία μας ε, θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στην χρήση νέων τεχνολογιών, τονίζοντας το ρόλο αυτών των νέων τεχνολογιών σχετικά και τη σχέση που έχουν συγκεκριμένα με την ελευθερία έκφραση. Επίση, διοργανώσαμε ένα σεμινάριο τον Οκτώβρη στην Βαρσοβία, στα πλαίσια του ΑΣΑ. Και ε, και στην Αίγυπτο διοργανώθηκε επίσης ε, πριν από λίγο καιρό μία συνεδρίαση σχετικά με τη διακυβέρνηση στο διαδίκτυο και την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με αυτά, Πρόεδρε, νομίζω κάναμε μία επισκόπηση των εργασιών της ΚΟΧΟΜ τους περασμένους μήνες. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε στη συνεδρίαση τον Νοέμβριο και ευχαριστώ την Υποεπιτροπή για τις ε, καλές ανταλλαγές ε, απόψεων που κάνουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά, Πρόεδρε, για την αγαστή μας συνεργασία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάμαρσκιολτ στη νέα αυτή κατάσταση όπου βρισκόμαστε και όπου σημειώνεται αλλαγή στον τρόπο συνεργασίας των θεσμικών οργάνων στη βάση της συνθήκης της Λισαβόνας, νομίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμο. Θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα ανθρωπίνα δικαιώματα με ευρύτερο τρόπο και αυτό, όπως είπα, θα, θα φανεί πολύ χρήσιμο. Θα δώσω το λόγο στην Ναταλία τώρα. που είναι επικεφαλής του Γραφείου Βρυξελών της Διεθνούς Αμνηστίας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε να έρθουμε να σας μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε λίγα σχόλια από πλευράς ε, Διεθνούς Αμνηστίας για το ε, δίκτυο. Είναι αληθές ότι είχαμε υψηλές προσδοκίες από την Σουηδική Προεδρία αναγνωρίζουμε ότι αντιμετώπισε προκλήσεις σημαντικές, πολλές αβεβαιότητες σχετικά και αβεβαιότητα σχετικά με τις ε, θεσμικές αλλαγές, Λισαβόνα ή όχι, η οικονομική κρίση, η αλλαγή του κλίματος, αλλά όλες αυτές οι προκλήσεις πρόσφεραν και ευκαιρίες για να επανεπιβεβαιώσουμε για παράδειγμα, που τοποθετεί τι αξίε τη για τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν αυτά τα πράγματα να μπουν σε πράξη. Και γι' αυτό το λόγο ε, υποβάλαμε συστάσει προ την Σουηδική Προεδρία για να μεταφερθούν από λόγια σε πράξει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη συνολική διάρκεια τη Προεδρία στο επίπεδο του business as usual, η Σουηδική Προεδρία τα πήγε καλά συνέχισε να εργάζεται επί των κατευθυντήριων γραμμών, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπήρξε και ένας τομέας όπου η Σουηδική Προεδρία κατέβαλε ε, έξτρα προσπάθεια την οποία αναγνωρίζουμε σε ό,τι αφορά δηλαδή, την διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά και σε πρόσωπα. Ε, δημοσίευε την ατζέντα πριν από σχεδόν κάθε συνεδρίαση έκανε πολλές διαβουλεύσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επίσης δημοσίευσε το ποιο είναι υπεύθυνο για ποιο πράγμα. Και αυτό το αναγνωρίζουμε και προώθησε επίσης και την υπευθυνότητα των θεσμικών οργάνων. Γιατί ένα πρώτιστο καθήκον είναι βέβαια η πρόσβαση στις πληροφορίες. Ωστόσο, περιμέναμε περισσότερα. Περιμέναμε μια προώθηση των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών στο mainstreaming των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της Ένωσης, μιας συνέχειας, αλλά και τέλος στο θέμα της συμμετοχής. Και θα αναπτύξω λίγο αυτούς τους τρεις τομείς. Αναμέναμε λοιπόν να γίνει μια γνήσια προσπάθεια να ενταχθεί, να ενσωματωθεί, να γίνει το mainstreaming των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένα παραδείγματα. Έγινε επέκταση των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 17, αλλά υπήρχε και ένα πρόβλημα σε σχέση με τον περιορισμό των συζητήσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτά τα βήματα, σε αυτά τα φόρα, χωρί να ανέβει σε ένα επίπεδο παραπάνω. Αυτό το είδαμε στι σκέψει κορυφή με την Ινδία και τη Βραζιλία, όπου δεν εντάχθηκαν στην μερίσια διάταξη των συναντήσεων αυτών τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στη συνάντηση με την Κίνα επίση δεν περιλαμβάνεται. Και για τη Ρωσία, οι υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων ναι μεν περιλήφθηκαν στα speaking points της ε, Προεδρίας, αλλά δεν μπήκαν στα επίσημα έγγραφα της διάσκεψης, της τη. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλα πράγματα στους ε, τομείς αυτούς. Έγιναν κάποια θετικά βήματα και το υπενθυμίζουμε στους τομείς business and human rights στην κοινή δήλωση που έκανε η ε, Σουηδική Προεδρία και η μελλοντική Ισπανική Προεδρία μετά από την διάσκεψη αυτή και αναμένουμε και ορισμένα σημεία κλειδιά να περιληφθούν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Η βασική δηλαδή έννοια του καθήκοντος να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλο παράδειγμα της απόκλησης μεταξύ πολιτικής βούλησης και πραγματικών πολιτικών της Ένωσης και αυτό αναφέρεται βέβαια κυρίως στα εσωτερικά της Ένωσης αλλά πάντως αναφέρεται και στην ε, νομοθεσία των διακρίσεων. Αφενός βλέπουμε δηλαδή κάποια τολμηρά βήματα από τη Σουηδική Προεδρία όταν <coughs> επέκρινε για παράδειγμα τη νομοθεσία στην Λιθουανία κατά των ομοφιλοφίλων. Από την άλλη μεριά δεν είδαμε τέτοια δέσμευση στη συζήτηση του Συμβουλίου για τη νέα οδηγία όπου διαπιστώσαμε να υπάρχει μια έλλειψη ε, ηγεσία από πλευρά Σουηδικής Προεδρία σε άλλα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν και εσωτερική και εξωτερική διάσταση και ορισμένων που είχαν μπει και στο πρόγραμμα Στοκχόλμης. Για το δεύτερο μείζον θέμα, την πραγματική δηλαδή συνέχεια και συνεκτικότητα της, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούσε τον αποκλεισμό όπλων για τον Ουσπεκιστάν οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε το εμπάργκο αυτό θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί και όχι να υπαχθούν στα εθνικά συμφέροντα. Και ναι, μεν υπάρχει εντατικοποίηση του διαλόγου, αλλά παρόλα αυτά η εξοπιστία έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Άλλο παράδειγμα, τα βασανιστήρια. Ναι, μεν η Προεδρία κατέβαλε προσπάθειες, έθεσε ορισμένες θέματα, ορισμένες υποθέσεις βασανιστήριων, αλλά υπήρχε η ευκαιρία να προσεγγιστούν τα βασανιστήρια με συνολικό τρόπο και εσωτερικά και εξωτερικά. Για εσωτερικά είδαμε κάποια πρόοδο, είδαμε δηλαδή για τις ε, έκτακτες ε, απελάσεις, τις έκτακτες εκδόσεις κλπ. Αλλά άλλα πράγματα δεν θίγησαν καθόλου. Ένα θετικό παράδειγμα ήταν η συνένεση για τη δημοκρατία. Ήταν καλή αυτή η συζήτηση που επέτρεψε να δούμε ποια, ποιος είναι ο αντίκτυπος των διαφόρων μηχανισμών στην κοινωνία των πολιτών. Στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε περισσότερους μηχανισμούς. Χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση των υφισταμένων μηχανισμών. Για την Eastern Partnership είδαμε να συμμετέχουν περισσότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κάτι που επέτρεψε να έρθουν στο προσκήνιο τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως πρόκειται για μια διαδικασία. Ακόμα δεν έχουμε δει τα επίσημα έγγραφα που θα περιλαμβάνουν τα πράγματα αυτά. Τρίτος τομέας, η συμμετοχή. Η γνήσια διαβούλευση ξεπερνά, η γνήσια συνεργασία ξεπερνά τα πλαίσια της απλής διαβούλευση και ιδίω με οργανώσεις όπως η Αμνηστία. Ε, δεν πρέπει μόνο να είναι η Προεδρία έτοιμη να ακούσει και απαντήσεις, να δώσει feedback. Πρόκειται λοιπόν για μια αμφίδρομη σχέση και όχι απλώς παροχή πληροφοριών. Αυτή η πραγματική συμμετοχή δεν επετεύχθη, για παράδειγμα, στην αξιολόγηση του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, όπου οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ναι μεν ενημερώθηκαν, δεν έλαβαν όμως κανένα είδου feedback, ακόμα και αν είπαν ότι πρόκειται να μα βάλουν μέσα στην έκθεση. Το άλλο που θέλω να πω είναι ορισμένα συγκεκριμένα θέματα που είδαμε στον διάλογο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είδαμε να διαγράφεται μια θετική τάση προόδου στον ίδιο το μηχανισμό δηλαδή του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε να αντιμετωπίσει χώρες με τις οποίες έχει καλές σχέσεις και είδαμε ξεκάθαρες προτάσεις, συστάσεις, ε, χρονοδιαγράμματα όπως Γεωργία, Καζακστάν, Τατζικιστάν. Είδαμε όμως από την άλλη μεριά πολύ λίγη πρόοδο στον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια απλή ανταλλαγή απόψεων περισσότερο με χώρες όπως Ουσμπικιστάν, Κυρκυζιστάν και Ρωσία. Μία δυνατότητα πρόοδο εδώ είναι να γίνει μια συμφωνία με ορισμένε χώρε με την υπόθεση ότι αν δεν, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα ταμπού, ότι όλα θα μπορούν να τεθούν στην ε, ημερήσια διάταξη ανα πάσα στιγμή. Δηλαδή δεν αποφεύγουμε τα δύσκολα θέματα, μπορούμε να ρίξουμε όμως και ενδιαφέρον σε ορισμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Να μην υπάρχουν ταμπού λοιπόν, ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε θέματα κοινού ενδιαφέροντο και με τρίτες χώρες. Για τις κατευθύνσεις γραμμές διαπιστώνουμε θετική πρόοδο και κυρίως ε, στην συνεργασία με τι πρωτεύουσε και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις βασανιστήριων και στο διεθνές επίπεδο και στην ανταπόκριση από το ε, στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και για την προπαρασκευή του ε, Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για την χρήση των συστάσεων του UPR και ούτω καθεξής. Για να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με λίγα σχόλια ατενίζοντας την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία και εμείς θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε την Ισπανική Προεδρία να αναλάβει κάποια από την κληρονομιά της Φιδικής να συνεχίσει τις πρακτικές διαφάνειες που επενέσαμε στην αρχή της ομιλίας μας και να τις κάνει στάνταρντ, να τις θεσμοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα τη δημοσίευση των πληροφοριών, το οποίο κάνει τι, την ευρεία διαβούλευση που να ξεπερνάει και τα όρια της διαβούλευσης και να σημαίνει πραγματική συμμετοχή. Για τις κατευθυντήρες γραμμές ασφαλώς χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για να στερεοποιηθεί η πρόοδος που έχει γίνει σε κάθε επίπεδο. Ενθαρρύνουμε την Ισπανική Προεδρία να αρχίσει τη διαδικασία για την προσχώρηση στη Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι ένα βήμα που πρέπει να γίνει. Και ε, τώρα για τον ηγετικό ρόλο της ε, Προεδρίας. Είδαμε σε ορισμένες περιπτώσεις της Σουηδικής Προεδρίας και ανησυχού, ανησυχούμε λίγο. Είδαμε να λέει ότι ναι, ε, συμφωνούμε με αυτά που λέτε εσείς ε, σε Διεθνή Αμνηστία, αλλά ως Προεδρία δεν έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε τα θέματα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι η Προεδρία έχει και λόγο και ικανότητα και δικαίωμα και καθήκον να θέσει ορισμένα θέματα. Βεβαίω, έστω και αν δεν μπορεί να τα επιβάλλει. Αυτά θα ήθελα να πω και σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Αλόνσο. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε όντως χρήσιμους μηχανισμούς που όμως δεν εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο. Και αυτό είναι και ένα, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που ανέφερε η κυρία όλοι ότι υπήρξε δηλαδή από τους πιο φιλόδοξους στόχους της Σουηδικής Προεδρίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ομπιόλς, ο οποίος έχει συντάξει την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχε λάβει και τον λόγο όταν εντάμβανε η Ισραηλική Προεδρία. Κύριε Όμπιολ, θα θέλαμε να ακούσουμε σχόλια για την διάσκεψη της Μαδρίτης, γιατί περνάμε τώρα από τη Σουηδική στην Ισπανική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάθε φορά που αρχίζει ένα νέο εξάμεινο Προεδρίας, υπάρχει μια διπλή όθηση. Δηλαδή, η απόλυτα νόμιμη βούληση μιας κυβέρνησης που θέλει να σφραγίσει το εξάμεινό και από την άλλη η υπευθυνότητα που απαιτεί να υπάρχει μία συνέχεια από τη μία προεδρία στην άλλη. Εγώ όπως και εσείς κυρία Πρόεδρε πιστεύω ότι ο διορισμός της κυρίας ε, Άστον ε, ως ε, είπα του αρμοστή θα εγγυθεί όλη αυτή τη διαδικασία προχωρήματος. Εγώ Εγώ τα είχα πει και την προηγούμενη φορά και οι εκτιμήσεις μου για τη Σουηδική Προεδρία παραμένουν οι ίδιες. Ήταν μια πολύ σοβαρή Προεδρία και συνέβαλε στο να παραμείνουν σε κεντρικό σημείο των συζητήσεων και των προβλημάτων που απασχόλησαν το Συμβούλιο της Ένωσης στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς είχαμε μία συνεδρίαση μια μισή σε εκπρόσωποι δηλαδή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ισπανικής Προεδρίας και μας εγγύθηκαν ότι η πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συνεχίσει με τη γραμμή που ακολούθησε η Σουηδική Προεδρία. Η συνεδρίαση όπως γνωρίζετε κυρία Πρόεδρε δεν ήταν μια συνεδρίαση ειδική για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μορατίνος, την Κάρμεν την Υπουργό Άμυνας, τον, τον Υφυπουργό για την Ένωση Διέγκο Ρεγαρίδο και άλλους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο τώρα να σας ε, αναφέρω εδώ μια περίληψη της ε, συζήτησης. Φαντάζομαι ότι άμα είχε κρατήσει συνεδρία σε άλλη μια μισή μέρα θα είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου, αλλά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Εμείς ε, συγκεντρώσαμε την προσοχή μας σε διάφορα θέματα. λοιπόν, που είχαν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα τα αναφέρω και θα σχολιάσω σύντομα δύο από αυτά τα οποία τα θεωρώ κατεπίγοντα και αν όχι κατεπήγοντα πολύ σημαντικά. Μιλήσαμε για μία αξιοποίηση και βελτίωση στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας των υπερατλαντικών σχέσεων, όπως δηλαδή καλύτερες, πιο στενές σχέσεις με τη δίκηση Ομπάμα, Αναφέραμε κατά το εξάμεινο της Ισπανικής Προεδρίας ε, την πιθανότητα μιας διάσκεψης κορυφής με τις Ηνωμένε Πολιτείες και συζητήσαμε για θεσμοθέτησή τους, όπως γίνεται και με τη Ρωσία, δηλαδή να έχουμε δύο διασκέψεις κορυφής με τις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Να υπάρχει δηλαδή το και στο mainstreaming να είναι και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, μίλησαμε για τη σύσφυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής. Θα αναφέρω την Κούβα, που επίσης απασχόλησε εν μέρη της συζητήσεις μας. και τόσο οι εκπρόσωποι της Ισπανικής κυβέρνησης όσο και οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου διαπιστώσαμε ότι μετά από την αλλαγή αρχηγίας στην κουβανική κυβέρνηση υπάρχει μια σαφής βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλήσαμε για το Αφγανιστάν. υπάρχει κοινή ανησυχία για μια κατάσταση που δεν βελτιώνεται και, μια στρατηγική για την πολιτική βοήθεια και την ε, επισητιστική βοήθεια μπορεί να δώσει μία νέα όθηση στη χώρα. Να σταθώ όμως στα δύο θέματα που εγώ θεωρώ πιο σημαντικά από όλα και που θα έπρεπε να τραβήξουν την προσοχή της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά την Ισπανική Προεδρία θα γίνουν και τα πρώτα βήματα για τη λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης Ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για την πιο ενδιαφέρουσα και καινοτόμο πτυχή της συνθήκης της Λισαβόνας. Αλλά για να βρίσκεται και η πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο αυτών των πρώτων βημάτων που θα σφραγίσουν τη δράση της, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, ε, πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα στην υποεπιτροπή μας. Υπάρχει και μια δεύτερη ενδιαφέρουσα πτυχή συγκυριακά βέβαια. Στην Μεσόγειο υπάρχει ένα πρόβλημα αντίληψης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν τα λαμβάνει νομίζω πολύ σοβαρά υπόψη της ε, ή δεν τα εξετάζει κατά τον ίδιο τρόπο όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μία από τις μάστιγες των τελευταίων ετών ήταν, είναι η τρομοκρατία που έπληξαν δύο από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία και έχουμε και αυτό το θλιβερό θέαμα, το καθημερινά θλιβερό θέαμα ε, με τις ε, σχεδίες, τους λαθρομετανάστες, ε, όλους αυτούς που θαλασσοπνίγονται στη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1995 και μετά ανέπτυξε μια πολιτική συνεργασίας με τις όμορες μεσογειακές χώρες και στις οποίες έθετε το θέμα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως κεντρικό στοιχείο. Και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο διαπιστώσαμε όμως ότι αυτή, αυτό το θέμα ε, ήταν, αντιμετωπίστηκε αναποτελεσματικά. Και υπάρχει το εξής παράλογο. Είχαμε μία αποπολιτικοποίηση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ε, χώρες της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου όπου τελικά τα θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, καπελώθηκαν από ένα γενικότερο φουνξιοναλιστικό σχέδιο και από την άλλη μεριά εντελώς αντιφατικά Αμπλίμπιτουμ διαμορφώνεται μια νέου τύπου πολιτικοποίηση των σχέσεων με την συμπροεδρία. Και όλα αυτά ρυθμίζονται από τις Ισραηλοπαλαιστινιακές σχέσεις. Δείτε εσείς, η διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, διάσκεψη κορυφής, δεν έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπρόεδρο και έχει παραλύσει όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί όλα διέπονται από αυτές τις σχέσεις. Εχθές, ο Ισπανός, ο Γάλλος και ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκαν στο Παρίσι για να δουν πώς θα αποεγκλωβίσουν την κατάσταση. Αλλά είναι σημαντικό σε αυτή την Επιτροπή, όχι για γεωπολιτικούς λόγους, αλλά για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, τα θέματα ε, της ευρωπαϊκής Συνεργασίας θα πρέπει να συζητηθούν ενδετικά. Αυτό συζητήθηκε και στη Μαδρίτη, πρέπει να μας απασχολήσει και μας. Ε, είμαι σίγουρη ότι με την συνθήκη της Λισαβόνας ε, θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό οι εργασίες της υποεπιτροπής μας και θα ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ε, και οι εργασίες της ΚΟΧΟΜ ε, θα επηρεάσουν τις δικές μας εργασίες, όπως είπε και η κυρία Χάμασόλντ. Η Ισπανία είναι η τελευταία χώρα που θα αναλάβει την προεδρία της ΚΟΧΟΜ και θα μπορούσατε ίσως να ε, μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Τώρα, στον κατάλογο των ομιλητών, ο κύριος Πρωτεσέβιτς και ίσως ο κύριος Χάουιτ, μπορούν να μας μιλήσουν για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πώς οι εργασίες ε, του ΟΗΕ συνδέονται με τα θέματα ε, που ε, ήταν οι προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτές τις σύντομες παρουσιάσεις. Με ικανοποίησε πάρα πολύ η σύνοψη αυτή που μας παρουσίασε η Σουηδή Υφυπουργός για το πρόγραμμα της Σουηδικής Προεδρίας. Ακόμη περισσότερο χάρηκα διότι άκουσα πως στόχος της Σουηδικής Προεδρίας είναι να έχει ρόλο παγκοσμίου παίκτη η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα κάνω όμως ε, κάποια σχετικά σχόλια. Λόγω αυτής της ε, παγκοσμίου στρατηγικής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση σε πολύ κοντινές μας χώρες, όπως η Λευκορωσία παραδείγματος χάρη. Ούτε καν αναφέρθηκε αυτή η χώρα σε αυτή την σύντομη παρουσίαση των εργασιών της Ειδικής Προεδρίας. Παρόλα αυτά, ε, όπως ξέρω γιατί ηγούμε της αντιπροσωπείας, ε, ε, της διμερούς αντιπροσωπείας, γνωρίζω την κατάσταση εκεί και την περασμένη εβδομάδα είχαμε εδώ στις Βρυξέλλες τον Αλεξάνδρου Μιλινκέβιτς που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποψήφιος για το, για το βραβείο Ζαχαρόφ που μας είπε ότι ε, έχουμε αντιφρονούντες που έχουν θεωρηθεί αντιφρονούντες, ε, δηλαδή αντρισίες συνείδησες, ε, συγγνώμη, από την την αμνηστία και κρατούνται ακόμη στην Λευκορωσία και το βλέπουμε στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύτηκε πριν από, ένα, πριν από μία εβδομάδα και δεν υπάρχει ελευθερία του συνέρχεστε για τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, και τους οργανισμούς προστασίας ε, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Βιέσνα ή ε, το Ίδρυμα Φινλανδολευκορυσικό Ίδρυμα Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είναι καταχωρημένοι οργανισμοί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο έστειλε επιστολή στον κύριο Μπίλτε, ανέφερε εκεί όλα αυτά τα ζητήματα πριν ε, από την διμερή συνάντηση που είχε με τον ε, ομολογό του και ούτε καν απάντηση δεν πήρα σε αυτή την επιστολή. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε τη θέση ε, σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας για να παίρνουμε απαντήσεις από την Προεδρία. Όχι βέβαια, δεν χρειαζόμαστε νέες συνθήκες για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Τρεις μήνες περίμενα την απάντηση και ούτε καν ξέρω αν στη συνάντηση με τον ομόλογό του ήγηρε αυτά τα ζητήματα ή αν ανησυχούν αυτά τα ζητήματα η Σουηδική Προεδρία. Τίποτα. Σιγή. Τι να πω, ε, είναι ντροπή ε, επίσης, ε, η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχουν προσκαλέσει την Λευκορωσία. Η τωρινή Σουηδική ε, κυβέρνηση που ασκεί και την Προεδρία εκπώνησε το πρόγραμμα για αυτήν την εταιρική σχέση χρησιμοποιώντας το λεγόμενο κινέζικο πρότυπο της δημοκρατίας. Και από ό,τι κατάλαβα, αυτοί που εργάζονται ε, για αυτή την ανατολική εταιρική σχέση, ε, ε, μας μιλούσαν για το κινέζικο πρότυπο εκδημοκρατισμού και οικονομίας, ε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δουλειά μας να προάγουμε αυτά τα μοντέλα εμείς. Νομίζω ότι οι τόσο κοντινοί μας γείτονοι δικαιούνται ελευθερία στις επιλογές που κάνουν. Σας ευχαριστούμε κύριε Ποτεσέβιτς. ως επικεφαλής ε, της ε, αποστολής ε, φυσικά είναι σημαντικό να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες της Προεδρίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που διοργανώσατε αυτή την συνεδρία στην περασμένη εβδομάδα όπως συζητήσαμε με τον Αλεξάνδρ Μιλβίτσε για όλα αυτά τα ζητήματα και άλλους συναδέλφους. Νομίζω ότι ήταν Εποφελής αυτή η συνεδρίαση, γιατί μπορέσαμε να συζητήσουμε το θέμα των βελτίστων ε, πρακτικών. Κύριε Χάουιτ, ε, από πλευράς Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ε, πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ήρθα με λίγη καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη από τη Σουηδική Προεδρία που δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την παρέμβαση. Πάντω με την κυρία Αντρική, όπως είπατε και εσεί κυρία Πρόεδρε, πήγαμε πριν από λίγε εβδομάδες να παρακολουθήσουμε, ε, να συναντηθούμε την Σουηδική Προεδρία, μπορέσαμε να συζητήσουμε και την συγχαίρω γιατί έκανε πραγματικά υπέροχη δουλειά. Δύο θέματα προκύπτουν, προέκυψαν μάλλον, ε, από την πρόσφατη επισκεψή μας στην Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Οι αυστηρές απόψεις που διατυπώνονται σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Έθνη θέματα γυναικών και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Αυτό είναι μία από τα, ένα από τα ισχυρά μας σημεία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πάντοτε υπάρχει γραφειοκρατική καθυστέρηση μέσα στην, στα Ηνωμένα Έθνη και προς τα εκεί κινείται. Και όλες οι οργανώσεις γυναικείων δικαιωμάτων λένε ότι πρέπει, μας ζητούν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προάγουμε τα θέματα αυτά και μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και ότι όλα αυτά θα είναι χρήσιμα. Θα ήθελα ε, να ακούσω αν η Προεδρεύουσα μπορεί να τοποθετηθεί επί του θέματος αυτού στα τελικά της σχόλια, στην απάντησή της. Θα δούμε τώρα ποιο θα ε, ακολουθήσει στα ύψιστα αυτά αξιώματα των ΗΕ. Θα τον υποστηρίξουμε. Θα υπάρχει όμως και μια νέα εποπτική επιτροπή στο επίπεδο των ΗΕ Εθνών για θέματα γυναικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών. Και πάλι για την Προεδρία τη Επιτροπή αυτή μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα και από ευρωπαϊκή πλευρά, να δούμε αν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια ευρωπαϊκή υποψηφιότητα. Πολύ ζωντανή ήταν επίση η συζήτηση, παρόλο που δεν θα συμφωνηθεί η αναδιάρθρωση του ε, αρμοδίου οργάνου των Εθνών μέχρι το 2012, αλλά και στην έκθεση της θα δούμε μια τρίτη επιτροπή με παγκόσμια αρμοδιότητα βασισμένη στη Νέα Υόρκη και μια για το Συμβούλιο βασισμένη στη Γενέβη και νομίζω ότι θα μπορεί να παίξει ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο. Πάντως η συζήτηση εξακολουθεί να διεξάγεται και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν, θα, αν πρόκειται να, ε, να προταθούν άλλα πράγματα σχετικά με αυτό. γιατί ακόμα υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Και δύο ακόμα θέματα εξωτερική πολιτική που είναι λιγότερο σχετικά, αλλά έχω δυνατότητα να σα θέσω ερωτήσει τώρα. Το άνοιγμα του γραφείου είναι μια ε, θαυμάσια εξέλιξη και αν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες που μπορείτε να δώσετε για το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τέλος, ένα θέμα το οποίο έφτιαξα εγώ στη Νέα Υόρκη και το επαναλαμβάνω εδώ σε σχέση με την έκθεση Gold Store. Ήταν τεράστια συζήτηση που έγινε και δικαίω και στην ακρόαση που έγινε στην Επιτροπή μας και στην Υποεπιτροπή μας φέτος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι για ότι η μεγαλύτερη ανησυχία που θα πρέπει να έχουμε είναι αν θα, μπορέσουμε, αν θα μπορέσουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνήσουν επί ενός κειμένου. Αυτό όμως δεν είναι το βασικό. Το βασικό είναι ότι διαπιστώνει μια έκθεση ότι έγιναν βαρύτατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγκρουση της ε, ζώνης της Γάζας και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι το θέμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν θα πρέπει εδώ να επιτυχθούμε ημέν κατά, κατά τον ΔΕΗ για τα όσα δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε, αλλά θα έπρεπε μάλλον να συνεργαστούμε επικοδομητικά και με το Ισραήλ και με του Παλαιστινίου και με τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να δούμε ώστε, ότι το ουσιώδε αυτό θέμα που θίγει η έκθεση θα ληφθεί εν τέλει υπόψη. Εγώ θεωρώ ότι τα τρία μέρη που αναφέρει η έκθεση θα αναλάβουν εν τέλει έρευνες και ότι θα τα ανταποκριθούν θετικά και επικοδομητικά στο κείμενο της εκθέσεως. Ήθελα να το πω αυτό και δημοσία και να θίξω και το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Ο Γκόλτστον, δικαστής, προσκλήθηκε στην Επιτροπή, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσέλθει για διαφόρους λόγους. Αυτό είναι ατυχές βέβαια, γιατί θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον για μας να μπορέσουμε να ακούσουμε τις παρατηρήσεις του από τον ίδιο. Δεν ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Γι' αυτό θα επανέλθω τώρα στην κυρία Έλινορ Χάμερσκιολτ και θα δώσω και στην κυρία Αλόνσο τη δυνατότητα να παρέμβει. Α, α, υπάρχει όμως μια βουλευτής. Πριν, πριν ακούσουμε την κυρία Χάμερσκιολτ, ας ακούσουμε την κυρία Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για τον Ταουφίκ Μπεμπρίκ, δημοσιογράφο και ποιητή από την Τινησία, ο οποίος καταδικάστηκε μέσα από περίεργες και θολές ε, κατηγορίες ε, για ποινικά ζητήματα που δεν ε, πείθουν κανέναν. Βλέπουμε λοιπόν τελευταία ένα κυνήγι κατά των προασπιστών, ε, άνευ προηγουμένου κατά των προασπιστών ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, την Ισία, αντίπεινα, περιορισμοί, κρατήσεις κλπ. και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο γενικής αδιαφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας εκπρόσωπος της Ένωσης και ή της Κομισιόν ήταν παρόν σε αυτήν την δίκη. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι εδώ για μη παροχή βοήθειας έχοντα κίνδυνο. Και σύμφωνα και με τις αμοιβαίε συμφωνίες και δεσμεύσεις που έχουμε με την, ε, την Ισία, είναι υποχρέωσή μας να θυμίσουμε του κυρίου Μπεναλή ότι όλα αυτά είναι αντίθετα με τις συμφωνίες. Και θα πρέπει να το ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τινησία σας ευχαριστούμε κυρία Κιλ Νίλσεν, ε, κυρία Χάμενχολ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω εν συντομία να απαντήσω στις ερωτήσεις που με απίθυναν τα μέλη της Υποεπιτροπής και να σχολιάσω και κάποιες από τις παρατηρήσεις ε, της κυρίας Αλόνσο. Επιτρέψτε μου να ζητήσω από την κυρία Νό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να σχολιάσει ε, τα ζητήματα, τα ερωτήματα που απευθύνονταν και προς την Προεδρία και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω με ένα ζήτημα εγκάρσιο που προέκυψε σε διάφορα από τα ερωτήματα δηλαδή το θέμα του mainstream, τη ένταξη του ζητήματο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκαν δύο διαστάσει του ζητήματο. Πρώτον, σε ποιο βαθμό συζητούμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε πολιτικό επίπεδο. Και δεύτερη διάσταση, η καθημερινή εργασία σε αυτό το τομέα τη ένταξη δηλαδή του θέματο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε τι πολιτικέ. Θα ήθελα απευθυνόμενοι στα μέλη της Υποεπιτροπής και σε όλους τους φορείς, τον, σε όλους τους περασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δούνε τα ανακοινοθέντα τύπου όλων των ε, διασκέψεων που έχουν γίνει και υπάρχει ε, πολύ διαθέσιμο, με, διαθέσιμο υλικό από όλες από όλα τα βήματα που έχει κάνει η Σουηδική Προεδρία. Έχουμε ε, γύρει το ζήτημα σε πολλά φόρα. η κοινή δήλωση, η σημερινή κοινή δήλωση, Φερρυπίν, μετά από την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, υπάρχει ένα συγκεκριμένο τμήμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Ε, Διάφοροι Σουηδοί Υπουργοί, όπως ίσως ξέρετε, έχουν ενημερώσει το Κοινοβουλίο για διάφορες διαστάσεις, ε, ε, για διάφορα για διάφορες προσπάθειες που έχει κάνει η Σουηδική Προεδρία σε διπλωματικό επίπεδο αλλά το καθήκον αυτό που πρέπει να επιτελέσουμε, το mainstreaming ε, και στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, είναι ένα θέμα που απασχόλησε την Προεδρία στην καθημερινή βάση. Ε, σας παραπέμπω στις δηλώσεις που δημοσιοποιούμε, σε δράσεις που αναλαμβάνουμε, παρότι δεν είναι όλες υπό την αιγίδα της COHOM ή στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της ΚΕΠΑ όταν ε, είμαστε στην Αλοδαπή, στις αποστολές που κάνουμε και την ενσωμάτωση του θέματος ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές. Φυσικά, επιδέχεται βελτιώσεις ε, η ε, στρατηγική μας, αλλά πάντως ενεργά προωθούμε αυτό το θέμα. Επίσης, ε, προσπαθούμε να τονώσουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κοινότητα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βερξέλλης και την Πολιτική Επιτροπή και Επιτροπή Ασφαλείας. Προσπαθούμε να εμπλέξουμε όλες τις κυβερνητικέ οργανώσεις στο έργο μας. Τώρα, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Πατασέφιτς ε, για τη Λευκορωσία. Ε, αληθεύει ότι δεν αναφέρθηκα σε αυτή τη χώρα ρητά, κυρίως ε, διότι είναι... από τις χώρες με την οποία είχαμε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως ε, μας έχει ούτως ή άλλως απασχολήσει η κατάσταση στη Λευκορωσία και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας τα πλαίσια ακριβώς των ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Έχουμε τα συμπεράσματα της 17ης Νοεμβρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημοσίευσε το Συμβούλιο και διάφορα άλλα που είπε ο κύριος ε, Ποτασέβιτς φυσικά αντιστοιχούν σε ανησυχίες ε, που έχουν, έχει εκφράσει ήδη το Συμβούλιο. Ε, θα ε, δώσω συνέχεια στο θέμα, θα δω τα επιμέρους ζητήματα που θίξατε στην επιστολή σας και θα σας στείλουμε απάντηση η κυρία Αρνό ίσως θέλει να σχολιάσει περαιτέρω αυτό που είπε ο κύριος Ομπιόλς ε, για τη Μεσόγειο. Εν συντομία εγώ να πω πως ε, υπάρχουν διάφορες μορφές ε, ανταλλαγών με τους γείτονες μας στη Μεσόγειο για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά ε, όπως τα εργαλεία που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ αυτό και συγκεκριμένο επίπεδο να κάνει ανταλλαγή εμπειριών. Πάω στα θέματα του ΟΗΕ τώρα που αναφέρθηκαν η αναθεώρηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΟΗΕ. Είναι βασική πρόκληση για τα ε, προσεχή χρόνια. Ε, αυτή η αναθεώρηση ε, γίνεται για ένα σχετικά νεότευτο όργανο και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις αρχικές αποφάσεις αυτού του οργάνου αρχίσαμε τις ανταλλαγές απόψεων ε, σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση και σχετικά με το ε, ε, τους στόχους που θα έπρεπε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να δείτε πόσο ανοιχτό πνεύμα έχουμε και πόσο δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, στο παρόν στάδιο ακούμε τις απόψεις όλων. Δεν υπάρχει κοινή θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση, γιατί ε, περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, των εταίρων μας που συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μας ε, να ακούσουμε ό,τι έχει σχέση με αυτή την αναθεώρηση πριν καταλήξουμε συγκεκριμένη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Κύριε Χάουιτ, ε, αναφερθήκατε σε αυτά που κάνουμε για να δώσουμε συνέχεια στην έκθεση Goldstone. μίλησα διεξοδικά για αυτό το θέμα. Όταν σας ενημέρωσα πριν από κάποιες εβδομάδες, επιβεβαιώνω σήμερα ότι ε, φυσικά αποδίδουμε τη δέουσα σοβαρότητα σε αυτή την έκθεση από πλευρά Ένωση και βασιζόμαστε στην ε, κοινή θέση ε, για την ανάγκη που υπάρχει για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ανάγκη να μπορεί να αποδοθεί ευθύνη για την παραβίασή του. Έχουμε διαπραγματευτεί το κείμενο, αλλά δυστυχώ δεν έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κοινή θέση Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω θα υπάρξει συνέχεια και φυσικά θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε προσπάθειές μας ε, σε αυτό το πλαίσιο. Επιτρέψτε μου τώρα να σχολιάσω αυτό που είπε η κυρία Κιλ Νίλσεν ε, ε, η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων στην Τινησία είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει συνένεση ε, ζητήσουμε τον κύριο Ιντινούς να διερευνήσει ε, την κατάσταση ε, και να επανέλθει, δηλαδή να κάνει εισηγήσει σε σχέση με τις κινήσεις που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μας απασχολεί ήδη το ζήτημα, το ερευνούμε. Θα ήθελα τώρα να ασχολιάσω ένα γενικότερο θέμα, δηλαδή η σχέση ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική εργασία μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Αλόνσο, κυρία Αλόνσο τον έφερε, αλλά ίσως θα μπορούσα να το συνδέσω με σχόλια που έκαναν άλλα μέλη της Υποεπιτροπής. Αναγνωρίζουμε ότι ε, είναι αλληλεσυμπληρούμενες οι δράσεις, αυτά που κάνουμε δηλαδή μέσα στα κράτη-μέλη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ικανότητα που έχουμε ως Ένωση να δράσουμε σε εξωτερικό επίπεδο. Έχουμε πλήρη επίγνωση της σχέσης. Ε, φυσικά μπορούμε να ε, τη βελτιώσουμε. Ε, και θα ήθελα να σταθώ ε, σε ε, δύο από τα ζητήματα που αναφέρετε. Δηλαδή, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό εντάσσεται πλήρω στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη και ο Υπουργό για τη Μετανάστευση μίλησαν την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Είναι ξεκάθαρο το υποστηρίζουμε. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και γι' αυτό ανεβάζουμε το υλικό στην ιστοσελίδα μα. Υπάρχει και ένα κομμάτι για τα θεμελιώδη δικαιώματα και όλα τα στα ζητήματα για την προστασία δηλαδή των πολιτών και ε, είναι ε, ξεκάθαρο το λαμβάνουμε υπόψη στα πλαίσια των εργασιών για την οδηγία για την κατάργηση της ε, διακριτικής μεταχείρισης. Θα ήθελα επίσης να κάνω άλλες δύο σύντομες παρατηρήσεις. Η κυρία Αρνό μπορεί να, και η εκπρόσωπος του είπατε προς όπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να σχολιάσουν περαιτέρω αυτό το θέμα. Τέλο πάντων, ε, ήθελα να μιλήσω για την αλληλεπίδραση, για τη διαχείριση των κρίσεων, για την αναπτυξιακή βοήθεια ανάμεσα στι δικέ μα εργασίε και εργασίε όλων. Ε, και συγκεκριμένα να μιλήσω για τα πρότυπα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ καλύτερο να έχουμε ένα γραφείο εδώ στι Βρυξέλλε, σε μία επιτόπου εκπροσώπηση, γιατί έτσι θα συντονίζουμε καλύτερα τη δράση μα. Ε, η κυρία Αλόνσο τέλος, ε, Πρόεδρε, μας μίλησε για το feedback. Ε, και ότι θα ήθελε, θα επιθυμούσε καλύτερη ενημέρωση από πλευρά τη Ιουδική Προεδρία για τα όσα έχει κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα απαντήσω ω εξή. Πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα αυτό και καλό θα ήταν, εφόσον έχουμε ακόμη ένα μήνα, να κάνουμε ε, μετά την τελική ενημέρωση τη Υποεπιτροπή, γιατί μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση στο μεταξύ και ε, προσπαθούμε να έχουμε στενή σχέση με του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την κοινωνία των πολιτών, με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Επανώνουμε διαρκώ, αλλά ε, και φυσικά μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό που κάνουμε. Και αυτό το ζήτημα που έθεσε η Διεθνής Αμνηστία είναι γενικότερο και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια συνέχεια για την αξιολόγηση. Τώρα για την κατάσταση στην Κίνα θα έλεγα ότι ακόμη βρισκόμαστε σε ένα προώρο στάδιο. Αναγνωρίσαμε την σημασία να υπάρχει και ενημέρωση και αλληλεπίδραση με την κοινωνία των πολιτών και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας. Αλλά μόλις τώρα αρχίσαμε τη συζήτηση του θέματος της αξιολόγησης εν μέρη διότι ασχολούμασταν με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του τελευταίου γύρου ε, συζητήσεων με την Κίνα. Εν συντομία, Πρόεδρε, για αυτό το ζήτημα θα ε, σας ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστούμε, κυρία Χάμερσελτ. Θα θέλαμε να ακούσουμε και άλλα σχόλια. Μιλήσαμε πολύ για συνοχή και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει ένα σημείο που θα ήθελα να αναπτύξω για αυτά που μας ε, ανέφερε ο κύριος Χάουιτ ε, σχετικά με την επίσκεψή του στον ε, ΟΗΕ. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα των γυναικών, της ασφάλειας και της ειρήνης. Και εγώ στο, μέσα στα πλαίσια του δικού μου μικρόκοσμου θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε δύο επιτρόπους της απερχόμενης επιτροπής την ε, κυρία Φερέρα Βάλνερ και Γουόλστρομ που πρόθυσαν αυτά τα θέματα. Όπως είπε και η Λεωνόρ Χάμερσολτ, έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένες πρόοδοι μετά τον Δεκέμβριο για το θέμα ειρήνης ε, ε, γυναίκες και ασφάλεια. Υπάρχει ένα πάνελ σχετικά, ένα training συγγνώμη, αλλά υπάρχει και ένα άλλο training ε, που αφορά στην αστική συνεργασία και στην πολιτική βοήθεια. Τον Οκτώβριο η Σουηδική Προεδρία κάλεσε ε, τα κράτη-μέλη για να τους ρωτήσει ε, στα πλαίσια της 13, του 1325 ψηφίσματος ποια ήταν η θέση τους και τι έχουν κάνει για τις γυναίκες, την ασφάλεια και τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών ειρήνης. Και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει γιατί του χρόνου θα θέλαμε να γίνει μια ε, αναθεωρητική διάσκεψη για αυτό το ψήφισμα. Ο κύριος Χόουιτ είπε ότι υπάρχουν πρόοδοι στον ΟΗΕ που πρέπει να ενθαρρύνουμε. Η όλη δομή όμως πρέπει να προχωρήσει στους επόμενους μήνες, διότι πάντα υπάρχει το ρίσκο. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να διοριστεί ένας ειδικό εισηγητής για το θέμα της βίας στους πολέμους και έχουμε 16 χώρες της Ευρωπαϊκής, τη, συγγνώμη, του ΟΗΕ μόνο που έχουν ένα εθνικό σχέδιο και μόνο τρεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τους 27, ε, απ, έξω έχουμε τρεις Αφρικές, ε, αφρικανικές χώρες, μία Λατινοαμερικανική και την Ορβηγία που έχουν ένα τέτοιο πρόγραμμα σε όλους τους ε, εταίρους μας θα πρέπει να πιέσουμε και στις χώρες του Μαγκρέμπ ε, και της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικανικής Ένωσης. Τώρα εγώ δεν ξέρω αυτό το Overseeing Committee που ανέφερε ο κύριος Χάουιτ, αλλά θα, θα μπορούσα να ενημερωθώ και να, να, να, δω τι γίνεται. Για... Α, α, λέει Μιλήτρια. Για το θέμα του κυρίου Ομπιόρης για την Μεσόγειο. Μα για το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόοδου πρόκειται λοιπόν για μια ιδιαίτερα κριτική περιοχή. Ε, ξέρετε ότι όλα επικεντρώνονται γύρω από την Ισραηλο-Παλαιστινιακή κρίση. Συμφωνούμε όμως ότι πρόκειται για μία ζώνη με ιδιαιτερότητες ε, ε, και με μία ζώνη με προβλήματα. Ε, πρέπει να την παρακολουθήσουμε σίγουρα. Δεν λέω εγώ ότι δεν θα ήθελα να πάω, αλλά τέλος πάντων με όλες τις χώρες της περιοχής, εκτός από τη Συρία και τη Λιβύη, τη Λιβύη που δεν έχουμε συμφωνίες συνεργασίας, με την Τουρκία έχουμε τις ε, προδιαπραγματευτικές συμφωνίες. Έχουμε τέλος πάντων όλη αυτή την Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συναντιέται με όλες αυτές τις χώρες. Τώρα το κακό νέο είναι ότι στα πλαίσια της ε, συμφωνίας συνεργασίας η συνεδρίαση με την Τινησία ε, η συνεδρίαση έχει αναβληθεί. διότι μετά τις εκλογές η Τινήση που δεν ήταν και ιδιαίτερα ευτυχής με, με σχόλια που γίνανε σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέβαλαν αυτή τη συνεδρίαση. Πρέπει να το πούμε αυτό σίγουρα. Εμείς συνεχίζουμε όμως τις εργασίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνεχίζουμε το διάλογο με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Επιτροπή της Βενετίας επίσης κάνει τη δουλειά της, το Μαρόκο έχει προσχωρήσει σε συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εξελίσσονται τα πράγματα και στην Αίγυπτο. Μην πρέπει λοιπόν να βλέπουμε την κατάσταση ως ε, άσπρο μαύρο μόνο, ε, αλλά ε, υπάρχουν ε, δυνατότητες να συνεχίσει άνετα η συζήτησή μας στα πλαίσια των συμφωνιών μας. Και βέβαια υπάρχουν και μερικά πολιτικά ρίσκα τα οποία πρέπει να αποφύγουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το μόνο που ήθελα να πω επιπλέον είναι ότι η Σουηδική Προεδρία μας έδωσε την ευκαιρία να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε για το πώς συμφέρονται, συμπεριφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθηγητής Ιγκή, ο οποίος ε, είναι εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ και τον άκουσαν οι Ευρωπαίοι σε ένα workshop στη Στοκχόλμη, ε, ασχολείται με το θέμα της κοινωνικής ευθύνης για το οποίο μιλάμε εδώ και πολύ καιρό στην Ευρώπη. Και ε, πρέπει λοιπόν να ε, προβληματιστούμε για το πώς συμπεριφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα ζητήσουμε και μία μελέτη για να δούμε τι κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις στις τρίτες χώρες. Ελπίζω στα τέλη της επόμενης χρονιάς να τα έχουμε όλα αυτά και να το σκεφτούμε και για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Η κρίση τα βγάζει όλα αυτά στην επιφάνεια, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβληματιστεί ασχέτως κρίσεως. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε κυρία Αρνό. Η κυρία Χάμερ θέλει να κάνει μια δήλωση για το ψήφισμα 1325 ε, για την κατάσταση των γυναικών σε ενόπλη σειράξη. Καλά κατάλαβα, όχι. Είναι πολύ καλό που αναφέρθηκε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ... να δώσω το λόγο στην κυρία Χάμερσολντ Ε, για την εξωτερική διάσταση θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Για την εσωτερική και εξωτερική διάσταση, ε, ε, ξέρουμε ότι αναγνωρίζεται αυτό στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης και καλωσορίζουμε αυτή την κίνηση, αλλά σε ένα συγκεκριμένο τομέα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η σχέση της εσωτερικής και εξωτερικής δράσης, μετανάστευση προς το παρόν. Ε, πραγματευόμαστε αυτό το θέμα από πλευράς ασφαλείας και όχι από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το θέμα των συμφωνιών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες και θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην απεκδίεται τις ευθύνες που έχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή να υπάρξει επιστροφή αυτών των ατόμων χωρίς ε, να έχει, ε, έχουμε κατοχυρώσει, ε, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τη διαδικασία εξέτασης του ασυλού, το αν αυτό επιθυμούν ή να έχουμε κατοχυρώσει ότι δεν θα υποστούν κακοποίηση βασανιστήρια όταν επιστρέψουν στη χώρα τους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Ευχαριστούμε ε, κυρία Αλόνσο. Η σημερινή μας ε, συζήτηση ε, καλό θεμέλιο για την εκπόνηση της πολιτικής μας. Έχουμε ασχοληθεί με εκατοντάδες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάμερσολντ και την ε, κυρία Νόρντλαντ επίσης από πλευράς της Προεδρίας για τη συνεργασία μας ε, και είμαι σίγουρη ότι ε, θα αναλάβει άξια τη σκητάλη η Ισπανική Προεδρία και όλοι μας και από τα τρία θεσμικά όργανα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την ίδια πρόκληση και νομίζω ότι ότι αν συνεργαστούμε και συνεργαστούμε και με διεθνείς οργανισμούς θα μπορέσουμε να κάνουμε αποφασιστικές κινήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο για την ε, Τουρκία. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση κατά τις 5.30 και μετά και κλεισμένο των θυρών θα συζητήσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διαλόγου με την Αφρική, τη Ρωσία και την Κίνα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και θα γίνει εμπιστευτική παρουσίαση και κλεισμένων των θυρών για την κατάσταση σε αυτές τις χώρες ε, για να δούμε πόσο ο διάλογος αυτός μπορεί να ε, βελτιώσει την κατάσταση σε αυτές τις χώρες. Ε, λοιπόν, προχωρούμε τώρα στο πέμπτο σημείο της Μεσσίας Διατάξεως, Τουρκία. Παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση στην Τουρκία. Μόλις εξέδωσε έκθεση προόδου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε συνεδρίαση της Μεκτή Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, στις 26 και 27 Οκτωβρίου. Η κυρία Φλότ, ε, συναδελφός μας, ε, επικεφαλής αντιπροσωπεία στην Τουρκία, θα ξεκινήσει τη συζήτηση και έχουμε και την κυρία Μενεράιτεν που θα πάρει συνέχεια το λόγο γιατί είναι η συγγήτρια. Έχουμε τον κύριο που εκπροσωπεί ε, ε, ένα φορέα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και τον κύριο Γκάρνερ που είναι ε, ερευνητή και θα μιλήσει από πλευρά τη Διεθνού Αμνηστία. Έχουμε και τον κύριο Πιλάρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πρέσβη Σελίν Κούνεμα από την μόνιμη αντιπροσωπεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες και όλους ιδιαίτερα τον κύριο Πρέσβη. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Η κυρία Φλότχλ θα πάει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που ε, βάλατε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και η Κοπεχάγη στην Τουρκία είναι πολύ σημαντικά σημεία για την προσχώρηση. Και αυτό εμψυχώνει και τις ε, εργασίες της, ε, της ε, αντιπροσωπείας. Η, η τουρκική κοινωνία ζητά να γίνουν αυτές οι αλλαγές μεταρρυθμίσεις ε, που έγιναν στην Τουρκία γίνανε καταρχήν από τη λόγω εσωτερικής ζήτησης. Ε, η κοινωνία των πολιτών, ε, οργανώσεις, συνδικάτα, δημοσιογράφοι είναι αυτοί που απέτησαν να γίνουν οι αλλαγές. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία δημιουργούν πολύ έντονες τριβές και αυτό το διαπιστώνουμε και στα τελευταία γεγονότα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το κλείσιμο της, για για το προχώρημα της δημοκρατίας στην Τουρκία. Στις 13 Νοεμβρίου έγινε μία συζήτηση στην ε, Τουρκία όπου ο Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε να γίνουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις και ανέφερε και για την προπτική ενός νέου συντάγματος για την Τουρκία. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί από τους ε, Ευρωπαίους υπεύθυνους. Υπάρχει το κουρδικό, είναι ένα ουσιαστικότατο θέμα διότι αφορά και στην ελευθερία της έκφρασης ε, στην αστυνομοκρατία, στην εξουσία της, ε, του στρατού, όλα αυτά αλληλοσυνδέονται με το κουρδικό στην Τουρκία. Και το άνοιγμα αυτής της, δημοκρατικής, ε, της διαδικασίας συγγνώμη, εκδημοκρατισμού ε, είναι πολύ σημαντικό να συμβαδίζει και να αντιμετωπίζει μάλλον και το πρόβλημα των Κούρδων και στην πολιτική του και στην πολιτιστική του, κοινωνική του διάσταση αλλά και τη στρατιωτική του διάσταση γιατί υπάρχει και ένα θέμα αφοπλισμού ε, στις κουρδικές περιοχές και αυτό δημιουργεί διπολισμό σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο στην Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει την πρόκληση η Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποστηρίξει την δημιουργία μιας συνένεσης στην Τουρκία. Και η κυρία ε, ε, που έχει κάνει τη σχετική εισήγηση το τονίζει αυτό. Υπάρχει Επίσης ε, και το θέμα της δυνατότητα δυνατότητας ε, στην ε, Τουρκία, δικαίωμα απεργίας των υπαλλήλων, δικαίωμα του συναθρίζεστε, του συνεταιρίζεστε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά δικαιώματα. Και όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή οι αρχές εργοδοσία, εργαζόμενοι, συνδικάτα, έχουν καταφέρει να ε, ανοίξουν ένα δρόμο συζήτησης για να μπορέσουν να αρμονιστούν με τις ε, προδιαγραφές ε, της, της ΔΟΕ για τα κοινωνικά ζητήματα. Επίσης το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα που εφαρμόζεται πολύ πιο ελεγμένα και συγκρατημένα σήμερα μεν, αλλά συνεχίζει να υφίσταται. και ε, δεν καλύπτονται οι απαιτήσει ε, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή στον τρόπο εφαρμογής του 301. Και θα πρέπει να εγγυθούμε την ελευθεροτυπία και την ελεύθερη έκφραση. Αυτά είναι βασικά στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και Αυτά επίσης ε, προστίθενται και σε άλλα ζητήματα, ισότητα ανδρών γυναικών, κοινωνικές και πολιτιστικές πρακτικές που οδηγούν ας πούμε στον καταναγκαστικό γάμο ή στα εγκλήματα τιμής. Ε, Επίσης ελεύθερη έκφραση και τυπία είναι μίζωνα αιτήματα. Και στην έκθεση της Κομισιόν τονίζονται οι σχετικοί φόβοι για το πώς θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα η κυβέρνηση Ερντογάν. Για το θέμα της ε, κοινοτικής ε, Κοινοτική επανεισδοχής μεταξύ Τουρκίας και Ένωσης, γιατί το θέμα του ασύλου ας πούμε είναι ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει νομική βάση για να μπορεί κανείς να έχει διεθνή προστασία σε αυτή τη χώρα. Και οι συνθήκες κράτησης μπορούν πραγματικά να σε τραλάνουν. Δηλαδή, όταν χωρίς νομική βάση, χωρίς δυνατότητα προσφυγής κρατήσε και μάλιστα για ένα χρόνο που δεν μπορείς να ελέγξει πόσο θα είναι, ε, πρόκειται λοιπόν ε, πραγματικά για, για, για μια κατάσταση απάνθρωπη και υποβαθμιστική. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να τα, να τα προσέξουμε όλα αυτά ούτω ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των μεταναστών στην Τουρκία είτε ζητάνε άσυλο είτε όχι. Επίσης άλλες εκθέσεις μας μιλάνε για βία στα σύνορα. Λένε πολλές φορές ότι η Τουρκία είναι σουρωτήρη αλλά στα σύνορά της με τη Βουλγαρία και την ε, Ελλάδα ε, προχωρεί σε αστυνομικές επιχειρήσεις. Ελέγχει λοιπόν, μπορούμε εμείς να το δούμε δηλαδή τι γίνεται και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Και, αλλά όταν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται ε, είναι αρκετά αμφισβητούμενος. διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμεινε η Τουρκία να ξανασυζητήσει στις διαπραγματεύσεις αυτά τα ζητήματα. Επίσης, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ε, είναι αρκετά δραστήρια και έχει σημαντικές επιτυχίες. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί αυτήν την προσέγγιση μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα η Τουρκία να συνδιαλέγεται σε περιφερειακό επίπεδο, διατηρεί το διάλογο με όλες άλλες χώρες της περιοχής, Ισραήλ, Συρία. Υπάρχει βέβαια το Κυπριακό. Και το πρωτόκολλο της Άγκυρας από τη μια όπου ζητούμε από την Τουρκία να σεβαστεί τις ε, δεσμεύσεις που ανέλαβε είναι πολύ σοβαρό και νόμιμο, αλλά ταυτόχρονα όλα θα πρέπει να αναλυφθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτω ώστε μία συμφωνία να ολοκληρωθεί στην Κύπρο στο εγγύς μέλλον και η συμφωνία αυτή να είναι ολοκληρωμένη και οριστική. Διότι σε όλο το Κυπριακό υπάρχει και ένα, ε, μια πρόκληση που είναι εσωτερική υπόθεση της Ευρώπης. Πρόκειται για μια εσωτερική σύγκρουσα στην Ευρώπη. Δηλαδή μπλέκονται εδώ πέρα μέσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Έθνη ως διαπραγματευτές όλη αυτήν την ιστορία. Πρέπει λοιπόν εμείς να υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται εξαφωτέρων των μερών για να έχουμε μία ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση για όλα τα σημεία, διότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο χωλαίνει σημαντικά τη διαδικασία και το οποίο χειραγωγείται επίσης στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. Όλοι λοιπόν έχουν συμφέρον να έχουμε λοιπόν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και γρήγορη λύση. Σας ευχαριστούμε κυρία Φλότρο. Τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στην κυρία Όμεν που θα σχολιάσει το σχέδιο ψηφίσματος που θα συζητηθεί στην Επιτροπή αυτή την Τετάρτη. Κυρία Πρόεδρε, στα αγγλικά, κυρία Όμεν εγώ θα περιοριστώ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Συζητούμε εδώ αυτό το θέμα και τη σωστή στιγμή μάλιστα διότι την Τετάρτη το πρωί θα καταθέσω την έκθεσή μου στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών όμως θα συνεχίσω καλύτερα στα Ολλανδικά. Νομίζω ότι η σημαντικότερη εξέλιξη το πρόσφατο αυτό χρονικό διάστημα όπως άλλωστε εξήγησε η κυρία Φλότρα είναι η ευρεία συζήτηση που έχει αρχίσει τώρα στην Τουρκία για Κούρδους και Αλεβίτες. Εγώ νομίζω ότι έχει, έχουν γίνει σημαντικά και θαραλέα βήματα. Θαραλέες ανακοινώσεις και βέβαια αυτές τις ανακοινώσεις πρέπει να τις ακολουθήσουν και δεσμεύσει και από πλευρά Κοινοβουλίου και κυβερνήσεω. Εγώ πάντως θα ενθαρρύνω με την έκθεσή μου όλους τους θεσμούς στην Τουρκία και καθώς και την κοινωνία των πολιτών να συνεχίσουν στην πορεία αυτή. Αντιλαμβάνομαι τις έντονες ευαισθησίες στην χώρα αυτή, αλλά πρέπει να δηλώσουμε και εμείς σαφώς ότι το δημοκρατικό αυτό άνοιγμα είναι μια καλή αρχή, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Στην έκθεσή μου περιλαμβάνω ορισμένες παραγράφους όπου γράφω ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συλλογικών δικαιωμάτων γίνεται για αυτήν την ε, προστασία πρόβλεψη σε ένα αριθμό νόμων, αλλά οι νόμοι αυτοί δεν λειτουργούν πάντοτε. Διότι ακόμα λείπουν οι μηχανισμοί επιβολής. Και επίσης εξακολουθεί να υπάρχει μια εσφαλμένη νοοτροπία. Νοοτροπία ε, διακρίσεων κατά των γυναικών, κατά ορισμένων κοινωνικών στρωμάτων κλπ. Άρα λοιπόν και εδώ πρέπει να είναι ισχυρή η θέληση να αλλάξουν ε, ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά, σε αφορά τη σύναψη γάμου. Υπάρχουν νόμοι που δεν λειτουργούν πάντοτε. Θα τα ξαναπώ εγώ λοιπόν αυτά στην έκθεσή μου εκτός από την υλοποίηση, υπάρχει έλλειψη και κατάλληλου δικαστικού μηχανισμού. Υπάρχουν ελλείψεις στο δικαστικό μηχανισμό. Έχω ξαναπεί ότι η δικαιοσύνη στην ε, Τουρκία είναι μεν ανεξάρτητη, αλλά δεν είναι και ακομάτιστη πάντοτε και γι' αυτό έχει σημασία μεγάλη σημασία να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στον δικαστικό μηχανισμό. Αυτό θα πω και στην έκθεσή μου, ότι δηλαδή πολύ σύντομα θα πρέπει να ψηφιστούν νόμοι για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Ένα τρίτο θέμα είναι τα δικαιώματα των συνδικαλιστών. Διαπιστώσαμε και τελευταία μάλιστα ότι έγιναν απαγορεύσεις συνδικαλιστικών κινήσεων, απεργιών και άλλα, με δικαστικές αποφάσεις. Το ίδιο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εφόσον αποτύχουν οι συλλογικές, οι προσπάθειες δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα να ε, προχωρήσουν οι εργαζόμενοι σε απεργία. Αυτό είναι και το τελευταίο τους όπλο. Τέλος, η ελευθεροτυπία. Τα άρθρα 301 αλλά και άλλα της ποινική δικονομίας χρησιμοποιούνται ακόμη τώρα για να γίνουν διώξεις και εγκλήσεις σε φυλακές αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν ανεκτά μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία που υποτίθεται ότι επιδιώκει να γίνει η Τουρκία. Για την ελευθερία του τύπου και αναφέρομαι κυρίως στον Όμιλο Ντόγκαν που αναγκάστηκε να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο και που νομίζω ότι αυτό το πρόστιμο δεν έχει καμία, δεν καμία απολύτως αναλογία με τα όσα συνέβησαν. Το αληθινό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ενώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που διαθέτουν για να προωθήσουν τα συμφέροντά του, Υπάρχουν δηλαδή μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων που συναπαρτίζονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικοδομή, σε ε, ορυχεία κτλ. Αλλά έχουν και ε, μέσα ενημέρωση στη διάθεσή του για να προωθήσουν τα ειδικά τους συμφέροντα. Αυτά είναι με λίγα λόγια τα κυριότερα θέματα τα οποία επιθυμώ να θέσω εν προκειμένου. Και τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα θέσω την Δετάρτη. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Όμεν Ρόιτεν. Έχουμε βέβαια το προνόμιο να ακούσουμε σήμερα μια πρώτη επισκόπηση της εκθέσεώς σας. Και βέβαια. Τα όσα θα συζητήσουμε σήμερα εδώ ίσως έχουν κάποια επηρεάσουν κάπως και το τελικό κείμενο της εκθέσεως σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κ. Γκέρελε που ε, είναι στον Εθνικό Σύνδεσμο 131 Εφημερίδων και είναι και υπεύθυνο για το BIA που είναι ένα δίκτυο και για το project ελευθερίας του τύπου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ε, εγκάρδια πρόσκληση. Εμείς μπορέσαμε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης ε, στην Τουρκία όταν η αντιπροσωπεία σας πέρασε από την Κωνσταντινούπολη. Εμείς ε, πολλές φορές συζητήσαμε αυτό το πρόβλημα και τονίσαμε πόσο άσχημα και ε, η δικαιοσύνη στον τομέα αυτών. Σίγουρα η κυβέρνηση του Ερντογκάν από το 2002 και μετά έχει ξεκινήσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις για να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. για να υπεραμηθεί δηλαδή και του καθεστώτος του υποψηφίου της Τουρκίας, της υποψηφιότητας της Τουρκίας. Και η τροποποίησεις ε, του ε, ποινικού κώδικα στην Τουρκία και οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι έπληξαν την ελευθεροτυπία στην Τουρκία και δεν είναι μόνο αυτό στους ε, δημοσιογράφους αλλά στους διαφωνούντες, ε, στους εκδότες, στους συγγραφείς και στους απλούς πολίτες. Όταν η κυβέρνηση θέλησε να επαναπροσδιορίσει το 2005 το νέο ποινικό κώδικα. Οι δημοσιογράφοι είχαν διαδηλώσει μπροστά από το δικαστικό μέγαρο για να σημάνουν τον κόδωνα του κινδύνου. Εγώ δεν θέλω να σας αναφέρω για όλα τα άρθρα ένα, αλλά έχουμε καμιά τριαντεριά δια, διατάξεις ε, στον ε, τουρκικό ποινικό κώδικα που περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση και εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχει και το άρθρο 301 που όλοι το γνωρίζετε, διεθνώς έγινε σκάνδαλο. Και όταν ο Ορχάν Παμούκ το βραβείο Νόμπελ κατηγορήθηκε όταν ο Βραντίν Καϊτά δολοφονήθηκε διότι δέχτηκε τις υπερεθνικιστικές απειλές. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι περίπου 5.000 άτομα κατηγορήθηκαν στην Τουρκία στα πλαίσια του 301 ή του 159 ε, που ήταν το αντίστοιχο άρθρο του προηγούμενου κώδικα. Να μην σας αναφέρω άλλα άρθρα του κώδικα, αλλά ορίστε η Λεϊλά Σάνα ε, η υποψήφια του βραβείου Ζαχάροφ ε, για το 1995. Η περίπτωση της ε, απεικονίζει πολύ καλά ποιες είναι οι διάφορες ε, προσεγγίσεις του, των τουρκικών δικαστηρίων όταν μιλάμε για ένα ίδιο θέμα. Ας πούμε, για ένα δικαστήριο το να εκφράζεται κανείς ε, για υπέρ των Κούρδων μπορεί να ε, θεωρείται αδίκημα, για άλλους όχι. Είναι δύσκολο να μιλάει κανείς ε, για δημοκρατικά στάνταρτ στην ελευθεροτυπία και στην ελεύθερη έκφραση, διότι τέσσερα χρόνια μετά από την έγκριση του ποινικού κώδικα, του νέου ποινικού κώδικα, δεν υπάρχει σχετική νομολογία ούτε για το 301, ούτε για δικήματα που αφορούν στην παρότρινση για τα κηρύγματα μίσους και Παρόλες τις ε, τροποποίησεις που έχουν γίνει, έχουν γίνει τρεις-τέσσερις τροποποίησεις, αλλά καταλήγουμε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Ας πούμε για, για τους αντιτρομοκρατικούς νόμους. Ε, λοιπόν, κοιτάστε, άμα εσείς λέτε φιλιρινικά πράγματα στην Τουρκία, ρισκάρετε 7,5 χρόνια φυλακή. Ο, Ναχμούτ Τορουκάν, που είναι δημοσιογράφος της Μιλιέτ, ο οποίος κινδύνευσε να αναφέρει την άποψη ενός τελέχους του ΠΚΚ σχετικά με το δημοκρατικό άνοιγμα της κυβέρνησης τον πήγανε στα δικαστηρία βάσει του άρθρου 7 του αντιτρομοκρατικού νόμου που λέει ότι η προπαγάνδα για μια, υπέρ μιας τρομοκρατικής οργάνωσης απαγορεύεται. Αλλά στα πλαίσια της αξιολόγησης θα έλεγα ότι σε επίπεδο της, της πρακτικής της δικαιοσύνης υπάρχουν προβλήματα, της απόδοσης της δικαιοσύνης υπάρχουν προβλήματα, διότι Παρά τις προσπάθειες προσαρμογής που γίνονται, στην πράξη έχουμε πολλά προβλήματα. Ο κίνδυνος φυλάκησης των δημοσιογράφων είναι πολύ σοβαρός. Γίνονται διαβήματα ούτως ώστε να μην είναι πια τόσο χοντροειδείς και χοντροκομμένες οι συλλήψεις ε, των ε, δημοσιογράφων και των διαφωνούντων. Διότι στο παρελθόν, όταν συλλαμβάνανε τους δημοσιογράφους, ε, δεν τους δίνανε ούτε πρόστιμα, ούτε αναστολή τους βάζαν κατευθείαν στη φυλακή. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο, ο λανθάνων κίνδυνος φυλα, φυλάκισης. Επίσης η ατιμορρησία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην Τουρκία. οι εκπρόσωποι των οργάνων της ε, τάξεως ε, οι οποίοι κατηγορούνται για βιοπραγίες ε, κατά των δημοσιογράφων τη χάνουν πλήρους Οι διαδηλώσει της Πρωτομαγιάς του 2007 και του 2008 στην πόλη και αλλού στην Τουρκία Είναι πολύ ουσιαστικό λοιπόν η ιεραρχία της αστυνομίας να λάβει τα μέτρα της ούτως ώστε να μπορεί να τιμωρεί αυτές, αυτά τα αστυνομικά λάθη και τις παρεκτροπές. Διότι η ατιμορρησία μειώνει το, τον ίδιο το ρόλο και την σημασία και το έργο της αστυνομίας προς την κοινή γνώμη. Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Θα δώσουμε το λόγο στον πρέσβη και μετά θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους ομιλητές. Thank uh, um, Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να μπορώ να είμαι παρόν σήμερα και να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας σχετικά με την πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Προσωπικά θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι για την ευκαιρία να προσέλθω εδώ τρεις μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως ε, μόνιμος εκπρόσωπος ε, της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένω να μπορέσω να συνεργαστώ και με τους Ευρωβουλευτές και με την Επιτροπή σας και υποεπιτροπή σας στη διάρκεια της θητείας μου εδώ, διότι αντιλαμβάνομαι πλήρως, όπως και καθένας, το σημαντικό ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Τουρκίας. Όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός Εξωτερικών και Μεν Μπαούς, υφυπουργό εξωτερικών και επικεφαλή των διαπραγματεύσεων από πλευρά Τουρκία, θα συναντηθεί με τα μέλη τη Επιτροπή σε λίγε μέρε. Σα υπενθυμίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγικό στόχο τη Τουρκία εδώ και δεκαετίε. Κάθε κυβέρνηση που έχει αναλάβει καθήκοντα στα τελευταία 46 χρόνια από την αρχική συμφωνία συνθέσεως του 1963 έχει θέσει τον στόχο της εντάξεως ως ε, ένα από τους θεμελιώδεις λήθους της ως ε, θεμέλιους ε, της πολιτικής της. Δεν είναι απλός στόχος της εξωτερικής πολιτικής. Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία προσχώρησης, η διαδικασία πορείας προς την προσχώρηση είναι και σημαντική κινητήριος δύναμης για τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε επιτελέσει τα τελευταία χρόνια και για την ενίσχυση του δημοκρατικού μας συστήματος και τη βελτίωση της νομικής βάσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν αναλυφθεί μέχρι τώρα έχουν δημιουργήσει και νέα νοοτροπία και, νέα, ε, και νέο πολιτισμό, πολιτιστικό πολιτισμό στην Τουρκία. Οι αντιλήψεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν μετακινηθεί επίσης σημαντικά έχει μπει πλέον το άτομο στο κέντρο του ε, νομικού συστήματος, είτε πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες, για νέους ή για πλέον ηλικιωμένους. Όλοι οι άνθρωποι παίζουν το ρόλο τους, η δημοκρατία ενισχύεται, τα τουρκικά στάνταρ στους χώρους των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών βελτιώνονται διαρκώς. Αυτό αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ετήσιες εκθέσεις πρόοδου της, αλλά και στα διάφορα κείμενα που ε, εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο πρόσφατα στο ψήφισμά του για την στρατηγική της διεύρυνσης που ψηφίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένουμε βεβαίως με ανυπομονησία και την έκθεση της κυρίας Όμεν Ρόιτεν που ε, κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι η Τουρκία ικανοποιεί επαρκώς τα κριτήρια της Κοπενχάγης για ε, να προχωρήσουν οι συζητήσεις, για ε, προματεύσεις για την ένταξη. Συνοψίζοντας, έχουν γίνει ε, σημαντικές νομικές μεταρρυθμίσεις. Σε λίγο χρόνο τροποποιήθηκε το Σύνταγμα σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις από το 2001 και έχουν ψηφιστεί οκτώ δέσμες ε, μέτρων. Από, με, ένα, με ένα σύνολο 53 νόμων που εγκρίθηκαν και έχουν συνέπειες και στο αστικό δίκαιο και στο ποινικό δίκαιο και στο εταιρικό δίκαιο και στις ε, δικονομίες και ούτω καθεξής. Σημαντικές βελτιώσεις έγιναν στα άρθρα που αναφέρονται στα δικαιώματα των γυναικών και στον αστικό και στον ποινικό κώδικα. Έχουν εκδοθεί και εγκύκλοι για την εφαρμογή των νόμων αυτών. Στον χρόνο που με έχετε διαθέσει δεν θα προλάβω να επισέλθω σε λεπτομέρειες αυτής της ε, σημαντικής διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, αλλά θα σημειώσω λίγες σημαντικές αλλαγές. Από το 2001, για παράδειγμα, καταργήθηκε η θανατική ποινή. Και αυτό μάλιστα, μάλιστα ενώ η Τουρκία υφίστατο μια βάρβαρη τρομοκρατική εκστρατεία. Έχουν γίνει και άλλες σημαντικές αλλαγές για την ε, καταπολέμηση των, ε, των βασανιστήριων και έχει εγκριθεί μια πολιτική της μηδενικής ανοχής, επίσης για την διδασκαλία και, τις, και την εξαγωγή εκπομπών σε διαλέκτους άλλες πλην της τουρκικής γλώσσας. Έχουν δοθεί λοιπόν η δυνατότητα επανεξέτασης καταδικών ε, στην ε, βάση των αποφάσεων που έχει ε, εκδώσει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, νομικές διατάξεις που εκδόθηκαν για θέματα ισότητας των φύλων και άλλα. Πρόσφατα η τροποποίηση του άρθρου 90 του συντάγματος διεθνείς συμφωνίες ε, στον χώρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπου τώρα υπερτερούν οι διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Τουρκία απέναντι στους εθνικούς νόμους. Έχει αλλάξει και η νοοτροπία, όπως είπα, και τομείς που μέχρι τώρα είχαν παραγνωριστεί, όπως τα δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, έχουν τώρα προχωρήσει στο προσκήνιο. Έχουν δημιουργηθεί θεσμοί για την επιβολή των σχετικών νομοθεσιών και αυτό έχει σαφώς θετική συνέπεια, θετική συνέπεια, θετικό αντίκτυπο. Για παράδειγμα, η νομοθεσία ε, για την καταπολέμηση των φόνων τιμής ή φόνων που οφείλονται σε παλές διαμάχες είναι πλέον γεγονός. Επίσης αντιμετωπίστηκε και το θέμα της ε, σχέσης μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, της προσαγωγής πολιτών ενώπιον των στρατοδικείων και για πρώτη φορά πριν από λίγα χρόνια ένας μη στρατιωτικός ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας, του Γενικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάζει θέματα αμυντικών δαπανών, είναι ε, υπό, τον πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο και το ανώτατο ε, Συμβούλιο Εκπαίδευσης. Εκεί έχουν αφαιρεθεί ορισμένοι περιορισμοί. Η επέκταση των πολιτιστικών δικαιωμάτων με την δυνατότητα που δόθηκε να διδάσκονται και άλλες διάλεκτοι πλήν της τουρκικής ήταν το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία η οποία συνεχίζεται, καθώς επίσης και ιδιωτικές, ε, ε ιδιωτική διδασκαλία των γνωστών αυτών σε, σε πόλεις όπως τα Άδανα και άλλες. Αλλά ορισμένα από τα σχολεία αυτά έχουν κλείσει λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος εκπομπές σε διάφορες γλώσσες και διαλέκτους, είναι δυνατές πλέον από το 2004. Οι περιορισμοί που επιβάλλονταν αρχικά έρονται τώρα, όπως θα σας εξηγήσω σε λίγο. Βέβαια, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι ένα σημαντικό στοιχείο και απαραίτητο τμήμα της προσπάθειας και για την εκπαίδευση το ίδιο και ε, εξαντλείται ο χρόνος μας. Πόσο χρόνο μου δίνετε ακόμη. Αν θέλετε παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Λυπούμε που δεν μπορώ να συνεχίσω την απαρίθμηση αυτών ε, των σημαντικών επιτευγμάτων, αλλά θα έρθω σε αυτά που ήθελα να τονίσω, που είναι με λίγα λόγια ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ε, είναι, βαίνουν σε ιδιαίτερο βάθος, η εφαρμογή, τους, η εφαρμογή υλοποίησή τους εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και πολλά έγιναν. Δεν θα έχουμε χρόνο για τους συναδέλφους. Μου δίνετε δύο λεπτά. Όχι. Καλά. Δέκα λεπτά. Αυτό είναι όλο. Παρακαλώ πείτε το συμπέρασμά σας. Θα τελειώσω εν τη αυτή περιπτώση αναφερόμενος στη νέα διαδικασία μεταρρυθμίσεως που ανακοινώθηκε πρόσφατα, το δημοκρατικό άνοιγμα, τη διαδικασία δημοκρατικού ανοίγματο, που ε, πρόκειται να ολοκληρώσει και να ε, αναπτύξει ε, τα όσα έγιναν, τα όσα επιτέθηκαν μέχρι τώρα, ως τμήμα αυτής θα ιδρυθούν και έδρες κουρδικής γλώσσας στα πανεπιστήμια. Νέα επιτροπή για τον αγώνα κατά των διακρίσεων θα δημιουργηθεί θα δοθεί η δυνατότητα εκπομπής στην κουρδική και άλλες γλώσσες και διαλέκτους. Θα επεκταθεί και αυτή. Λοιπόν, πάρα πολύ. Παρακάλεσα να ολοκληρώσετε. Συνεχίζετε. Μπορείτε να μας αφήσετε την δήλωσή σας. Μία τελευταία πρόταση, μία τελευταία φράση με την αδειά σας κυρία Πρόεδρε. Όπως είπε και η Αφρότερ προηγουμένως, ε, είναι θέμα βεβαίως προκαλούνται σημαντικές συζητήσεις με όλες αυτές τις ε, ε, μεταρρυθμίσεις αναπτύσσονται διάφορες απόψεις και θα πρέπει να είναι κατανοητό ότι η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μία μέρα όπως και η Ρώμη δεν σε μία μόνη μέρα. Είμαι βέβαια ότι θα μπορέσετε να απαντήσετε και σε ερωτήσει των συναδέλφων μου. Πρώτη και Χάουιτ. Τώρα. Και μετά έρθει το συνάδελφο. Αλλά πολύ σύντομα. Έχω τώρα πολλού που ζητούν το λόγο. Θα περνάμε περισσότερο σε δύο λεπτά. Κύριε Χάουιτ. Συγγνώμη, δεν ήθελα να μιλήσω πριν τους προσκεκλημένους και ίσως και ε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι θέλουν να ακούσουν πρώτα τους προσκεκλημένους και μετά να μιλήσουμε. Ναι, βεβαίως, γι' αυτό οργανώσαμε και την ακρόαση. Οπότε προτείνω όμως να ακούσουμε τα μέλη της Υποεπιτροπή ε, και μετά να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τη Διεθνού Αμνηστία και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλιώ δεν θα μπορέσετε, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε. Μάλιστα. Ε, έτσι για καθοδήγηση ε, θα μπορούσατε να μας πείτε για πόσα λεφτά μπορούμε να μιλήσουμε. Πρώτος ο κύριος Πρόντι, δύο λεπτά. Εγώ ήθελα να κάνω μια γενική τοποθέτηση για την ε, σημασία την οποία προσδίδω στη διαπραγματεύση με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα πολύ σημαντική που μπορεί να συμβάλλει επίσης σημαντικά στην δράση μας στο πλαίσιο της ε, παγκόσμιας πολιτικής για την ειρήνη. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω πώς πως αυτή η τόσο μεγάλη σημασία της διαπραγμάτευσης παρερμηνεύθηκε πολλές φορές ε, αναφερόμενη ως σύγκρουση πολιτισμών ε, πολιτιστική σύγκρουση μεταξύ Δύσης ε, και Ανατολής, Ισλάμ και Δύσης. Το πρόβλημα δεν είναι όμως το, η σύγκρουση μεταξύ ε, Δύσης και Ισλάμ, αλλά τα ίδια τα προβλήματα μέσα στο Ισλάμ. Η, θρησκευτική ε, και πολιτικοκοινωνική διάσταση που δεν διαχωρίζονται. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να οδηγήσουμε ε, τα Ισλαμικά κράτη στο να προχωρήσουν σε αυτό το διαχωρισμό θρησκείας πολιτείας και να προχωρήσουν ε, στην επιλογή της λαϊκότητας. Διότι αλλιώς άμα κάνουμε αυτού του είδους τις διακρίσεις οι βάσεις μας θα είναι εντελώς λάθος. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σύντομος. Ο κύριος Χάουιτ τώρα. Πρόεδρε, χαίρομαι που η κυρία Φλότρα επέστρεψε στην υποεπιτροπή του και ηγείται και της αντιπροσωπείας και χαίρομαι που η κυρία Μενερόιτεν ε, έχει αναλάβει το θέμα γιατί συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη διάσταση και χαίρομαι που είστε εδώ και χαίρομαι επίσης που στην υποεπιτροπή μπορούμε να οργανώνουμε τέτοιες συζητήσεις για αυτό το θέμα. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Υποεπιτροπή εδώ και χρόνια ασχολείται με το θέμα της Τουρκίας και θα συνεχίσει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό να κάνουμε, να απευθύνουμε επικρίσεις, ναι αλλά στις επαφές μας να αναγνωρίζουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, γιατί αλλιώς θα στείλουμε πλημελή μηνύματα προς συναδέλφους μας και καλωσορίζω και τον πρέσβη ε, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις τώρα και θα ήθελα να λάβω απαντήσεις από τους προσκεκλημένους. Πρώτον, η νομοθεσία, ε, ε, έχουμε, υπάρχει κολυσιεργία για την νομοθεσία για τα συνδικάτα και ε, είναι προς συμφέρον όλων να προχωρήσουμε. αλλά ακριβώς ποια είναι η άποψη της κοινότητας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αυτή τη νομοθεσία επί τη βάση των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Και όπως είπε και η κυρία Φλότρ, ναι, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο για το άρθρο 301, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα. Ποιε δυνατότητε ε, κατάρτιση έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για του εισαγγελεί και γενικά τους φορείς του συστήματο απονομή δικαιοσύνης, ούτω ώστε να κατανοήσουν ε, πώ μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση σύμβαση, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα. Τρίτον, ε, για το κουρδικό θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συγχαρούμε την Τουρκία γιατί έχει κάνει σημαντικότατα βήματα. Βέβαια είναι σοβαρό το ζήτημα και πολύ μεγάλο και πολλοί μας λένε ότι θα ζητηθεί συνταγματική μεταρρύθμιση ούτως ώστε να γίνουν αλλαγές για να ε, προστατευθούν τα πολιτιστικά δικαιώματα των Κούρδων. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε, ομοθυμία δεν υπάρχει στα βασικά κόμματα της Τουρκίας ούτως ώστε να ε, προκύψει αυτή η συνταγματική μεταρρύθμιση. Τι μπορεί να γίνει ούτως ώστε όλα τα μεγάλα κόμματα ε, στην Τουρκία να καταλήξουν σε αυτή τη συνένεση που χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε κύριε Χάουιτ. Θα ήθελα να δω μαζί σας τον κατάλογο των ομιλητών ε, και σας παρακαλώ ε, να είστε ε, σύντομοι. Ήταν ο Χατζηγεωργίου Evans, και μετά τους δύο εμπειρογνώμονες μας, ο κύριος Τάνοκ. Ε, πρόεδρε, ε, δύο ζητήματα θα σχολιάσω. Πρώτον, υπάρχει η εσωτερική διάσταση, δηλαδή το ένομο σύστημα της Τουρκίας και συγκεκριμένα οι μεταρρυθμίσεις ε, ε, της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για δημοκρατία. Είδα στο Βρετανικό τύπο το Σαββατοκύριακο μία υπόθεση για έναν νομοφιλόφιλο, ανοιχτά ομοφιλόφιλο, ε, που δολοφονήθηκε από τον πατέρα του. Ε, ε, και παρόσα μα είπε ο πρέσβης ε, αναφέρεται ότι αυτά τα εγκλήματα τιμής δεν οδηγούν σε σοβαρές έρευνες από πλευράς της αστυνομίας ε, και όταν γίνεται δίκη τελικά οι αποφάσεις είναι για πολύ μικρές ποινές, συμβολικές ποινές και οι μη μουσουλμανικές θρησκευτικέ κοινότητες ε, βλέπουμε τα δικαιώματα τους δεν προστατεύονται. Έχουμε ακούσει παράπονα επίσης από χριστιανικές ε, ε, κοινότητες και έχουμε και το, την σχολή της Χάλκης που παραμένει κλειστή. Δεν έχει εγκριθεί το άνοιγμα της σχολής και γίνονται προσπάθειες τα τελευταία δέκα χρόνια αλλά απόφαση ακόμη δεν έχει ληφθεί και αυτό θα συνιστούσε μια πολύ πολύ σημαντική κίνηση, ε, κάτι παραπάνω από συμβολική κίνηση που θα δείχνει ότι θα επιτρέπεται η εκπαίδευση των ε, ε, Ορθόδοξων Ιερωμένων στην Τουρκία. Αλλά τέλο πάντων, θα ήθελα να σχολιάσω και ένα άλλο θέμα. Ο ρόλο τη Τουρκία στον κόσμο για τη διατήρηση των κοινών μα αξιών και να μιλήσω λίγο και για την συμμετοχή τη στην Ισλαμική διάσκεψη. Πριν από δύο εβδομάδε διοργανώθηκε η συνεδρίαση στην στην Κωνσταντινούπολη και προσκάλεσαν τον πρόεδρο Αχμεντινετζάντε που ε, παρευρέθη και ε, περιγράφηκε ως φίλος της χώρας. Ο κύριος Αχμεντινετζάντε έχει παραβιάσει διάφορα ψηφίσματα του ε, για την διάδοση των πυρηνικών όπλων. Θέλει να εξαφανίσει από προσώπου γης το Ισραήλ. Έχει επίσης μιλήσει για το κρέμος με τον ομοφυλοφίλων από γερανούς προς δημόσια θέα Οπότε ένα τέτοιο άτομο πώς ακριβώς ταιριάζει με την ε, ε, ε, δεσμεύσεις της Τουρκίας και τη συνεισφορά της στη διατήρηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών. Ευχαριστούμε κύριε Τάνο και ζητώ συγγνώμη σας διακόπτω. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ αυστηρή γιατί είναι μακρύτερος ο κατάλογος των ομιλητών και δεν έχουμε χρόνο πλέον. Αν όλοι μιλάνε ε, ε, τρία λεπτά, δεν θα πρόβλημα, Θα ήθελα να ε, ρωτήσω κάτι τον πρέσβη σχετικά με το άνοιγμα της Τουρκίας και το κουρδικό ζήτημα. Έχετε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις αλλά ε, κατά τη γνώμη σας χρειάζεται μόνο τουρκική λύση. Δεν αναφέρθηκε στο διάλογο με τους ε, εκπρο... Ε, Κούρδους εκπροσώπους. Δηλαδή δεν αναγνωρίζετε το κουρδικό ε, ζήτημα και αν αυτό δεν γίνει πώς μπορεί να καταλήξετε σε μια θεμητή λύση. Ε, πρέπει να συζητηθεί το θέμα της συμμετοχής των Κούρδων στην κυβέρνηση, ή ε, το θέμα της ε, αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, που δεν συζητείται καθόλου και... ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, Κούρδοι πολιτικοί θύνοντες που είναι στη φυλακή. Χρειάζεται ένας ε, ανοιχτός διάλογος και μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να ρυθμιστεί το κουρδικό ζήτημα. Ε, ο προσκεκλημένος μας ε, αναφέρθηκε σε πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα ήθελα μία απάντηση από τον πρέσβη. Ευχαριστούμε, κυρία Ρέμπελς θα περιοριστούμε τώρα σε ένα λεπτό αν ομιλητή. Για τον εκπρόσωπο των δημοσιογράφων εδώ, θα βάλω μια επικεφαλίδα, επειδή προέρχομαι από την Κύπρο, εύκολα οι παριστάμενοι και ίσως και οι φίλοι από την Τουρκία να θεωρούν ότι αμέσως θα γίνει μια επίθεση. Θα προσπαθήσω να πω ότι θα είμαι αντικειμενικός και θα είμαι. Ήμουν στην Τουρκία, στην Μιχτή Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και παρακολούθησα επίσης πιο πρόσφατα μια δίκη στη Σμύρνη ενάντια σε 31 ε, Κούρδους συνδικαλιστές. Δεν υπάρχει το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων ούτε της απεργίας στους δημόσιους υπαλλήλους. Θέλω να ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια. Έχουν το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε, αλλά όχι το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της απεργίας. Οδηγήθηκαν σε δίκη με την κατηγορία ότι συμμετείχα στην οργάνωση μιας, παρακρα... μιας ε, τρομοκρατικής υποτίθεται οργάνωσης και η μόνη απόδειξη που προσήχθη ήταν τα εισιτήρια τα αεροπορικά που έδειχναν ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στον Τιάρπακυρ. Και βεβαίως παρακολούθηση ιδιωτική των τηλεφώνων και των email τους. Αυτό παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι το 301 δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι σήμερα το κοιτάζει με ένα διαφορετικό τρόπο η Τουρκία. Πρέπει να φύγει από το σύνταγμα αυτής της χώρας. Και κλείνω με το εξής, με ερώτηση. Έγινε μία δίκη ενάντια στο κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω πού κατέληξε αυτό το πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι εξακολουθεί να υφίσταται η δίκη αυτή. Μπήκε ένα πρόστιμο, αλλά υπάρχει ακόμα η κατηγορία της εισαγγελία ενάντια στο κυβερνόν κόμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω στον μόνιμο εκπρόσωπο της Τουρκίας. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχουν γίνει σημαντικές προοδοί στα, ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι αρκετά νέο. Εκείνο το οποίο δεν είναι νέο όμως είναι τα κείμενα. Τα οποία ερμηνεύουν αυτές τις πρόοδους. Λοιπόν, εσείς που έχετε μία εικόνα της ατμοσφαιρικής κατάστασης και της πολιτικής κατάστασης στη χώρα σας. Τι θα έπρεπε να γίνει ούτω ώστε να τονίσουμε αυτή την ενθαρρυντική πλευρά ε, στο προχώρημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας. Εγώ είμαι από χρόνια φίλος της Τουρκίας και υπάρχει μια τεράστια παρανόηση την οποία παραλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε ένα κοσμικό κράτος όπως η Τουρκία στα όρια της Ευρωπαϊκής Επίρου. Εάν δεν έχει κανείς κοσμικό κράτος στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άλλη ε, επιλογή που θα έχει η Τουρκία θα είναι να ασχοληθεί με το, με ότι βρίσκεται πίσω της. Όπου είχε μεγάλη επιρροή και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξεχνούμε τα ε, εξαιρετικά πράγματα που έκανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος εξυγχρόνισε την ε, Τουρκία, απελευθέρωσε τις γυναίκες. Και για κάποιο παράξενο λόγο οι Τούρκοι δεν μιλούν ποτέ για τα όσα επέτυχε ο Κιμολάτα Τούρκ. Oh. Eh, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον δημοσιογράφο, τον κύριο Ντέρογλου σχετικά με τις θρησκευτικέ ελευθερίες οι οποίες φαίνεται ότι συναντούν αρκετά προβλήματα στην Τουρκία παρά την πρόοδο που έχει γίνει και σχετικά με την επιστροφή των περιουσιών που έχουν κατασχεθεί από διάφορες μειονότητες. Πιστεύω, πιστεύει ότι είναι δυνατόν να γίνουν τα τελικά βήματα που χρειάζεται να γίνουν στα δύο αυτά ζητήματα. Επίσης το κοσμικό κράτος σε ποιο βαθμό μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει ε, μέχρι και στην τελευταία απομακρυσμένη περιοχή της Τουρκίας. Θεωρητικά υπάρχει παντού το κοσμικό κράτος, αλλά υπάρχει παραβίαση ελευθεριών για λόγους όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ε, ότι για λόγους τιμής υποτίθεται γίνονται διάφορα εγκλήματα. Σε ποιο βαθμό λοιπόν η προσαρμογή που γίνεται σε νομικό επίπεδο έχει αντίκρισμα και στο πρακτικό της μέρος, στην καθημερινότητα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γιαννάκου. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Άντρου Γκάρντερ να λάβει το λόγο πολύ σύντομα Δυστυχώ δεν είναι δυνατόν για παραπάνω από τρία λεπτά. Είμαι βεβαίω ωστόσο ότι θα μπορέσετε να περιοριστείτε στα πιο κεντρικά θέματα. Ε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι επίκαιρο το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Τουρκία ε, στα πλαίσια της συμφωνίας ανάμεσα στην Αρμενία και την Τουρκία. Όπως προαναφέρθηκε το άνοιγμα, το δημοκρατικό άνοιγμα της Τουρκίας για το κουρδικό, ίσως ε, ε, ε, ας δούμε αυτά τα, να δούμε αυτά τα δύο ζητήματα, τι σημαίνουν από ιστορικής πλευράς. τώρα βέβαια ακόμη συνιστούν ταμπού στην Τουρκία και θα ήταν καλό να προάγουμε πριν την ελευθερία έκφραση στην Τουρκία, γιατί τώρα όταν μιλάει κάποιο επικριτικά για το αρμενικό ή για το κουρδικό ζήτημα στην Τουρκία, δηλαδή δύο τομεί όπου ε, ε, εμποδίζεται η ελευθερία της έκφρασης ε, μέσω του ποινικού δικαίου το θέμα των ενόπλων δυνάμενων στην Τουρκία είναι ένα άλλο ζήτημα πέρα από τα πρώτα δύο που ανέφερα που οδηγεί συχνά σε ποινικέ διώξεις. Είναι σημαντικό μιλώντας για την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές ομάδες πληθυσμιακές που αποτελούν στόχο αυτών των ποινικών διώξεων. Όπως είπε ο κ. Σεντερογλου στην παρουσίασή του, ε, συχνά μιλάμε για δημοσιογράφους, για ακτιβιστές, ε, για εκδότες, για υπερασπιστές και δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για ακτιβιστές υπέρ των κουρδικών κομμάτων κτλ συνιστούν τον κατεξοχή στόχο το αυτών των ποινικών διώξεων ε, που παρεμποδίζουν την ελευθερία της έκφρασης. Τέλος πάντων, ε, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ε, ε, για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες στόχους, ε, νομίζω είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις διάφορες τάσεις ε, που σημειώνονται, δηλαδή τι είδους ομιλίες απαγορεύονται, παραδείγματο χαρή συχνά. Όταν συζητείται το θέμα της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία, ακούγεται η άποψη ότι ένας μικρός αριθμός άρθρων, συγκεκριμένα το 301 του ποινικού κώδικα, περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και ότι γενικότερα υπάρχει θέμα εφαρμογής εφαρμογής άλλων άρθρων. Ε, ε, δεν ευσταθεί αυτή η άποψη ε, σε ένα συγκεκριμένο βαθμό. Η εφαρμογή είναι σημαντικό πρόβλημα και θα επανέλθω σε αυτό, αλλά διάφορα θεμελιώδη προβλήματα που οδηγούν σε αυτές τις ποινικέ διώξεις που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης οφείλονται σε διάφορα άρθρα του ποινικού κώδικα που ε, αντιβαίνουν στο διεθνές ε, δίκαιο. Έχουμε το άρθρο 301, έχουμε και το άρθρο όμως 308 του ποινικού κώδικα. Το 308 ε, δεν επιτρέπει την πρόσβαση αυτών των ανθρώπων σε ένοπλες δυνάμεις. Να δύο συγκεκριμένα παραδείγματα άρθρων του ποινικού κώδικα που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης ε, υπάρχει και ένα γενικότερο ζήτημα της, το θέμα του περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης ε, και μην ξεχνάτε ότι σε επίπεδο διεθνούς δικαίου οι διατάξεις παρά είναι ασαφείς ε, και άρα δημιουργείται ένα είδος νομικού χάους που με τη σειρά του οδηγεί σε ποινικέ διώξεις. Τι να κάνω, θα σταματήσω κύριε Πρέσβη, βλέπετε ότι δεν είμαστε αυστηροί μόνο μαζί σας, αλλά και με τη Διεθνή Αμνηστία. Τα, ε, ακούστηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομος, σύντομος στις ε, απαντήσεις. Ε, θα σας δώσω δύο λεπτά για να είναι καλύτερο να είμαι συγκεκριμένη. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Δεν έχει ανάψει το μικρόφωνο το ο Πρέπει να επαναλάβω τώρα την πρώτη πρόταση που είπα. Λοιπόν, ε, εν συντομία να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους που έθεσαν ερωτήσεις ε, και χαίρομαι πολύ που σας συναντώ σήμερα. Ε, άκουσα συγκεκριμένα ερωτήματα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά που μπορούσα να σημειώσω για τις δολοφονίες. Το ζήτημα ρυθμίζεται από το νέο ποινικό κώδικα, αλλά χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστούν και οι δικαστέ ε, στις νέες νομοθετικές ε, ρυθμίσεις ε, και να αλλάξει η νοοτροπία των αστυνομικών αρχών, παραδείγματο χάρη, που διώκουν. Γι' αυτό και η κατάρτιση είναι είναι τον κάνει προϋπόθεση και γίνονται πολλά για να βελτιωθεί η κατάσταση θα ρυθμιστεί αυτό το πρόβλημα. Για τις μη μουσουλμανικές μειονότητες ε, έχει αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό διάλογος χάρη στο νέο νόμο ε, που ρυθμίζει το θέμα των περιουσιακών τους ε, στοιχείων. Για την σχολή στη Χάλκη είναι κοσμικό το τουρκικό κράτος και δεν προβλέπεται τέτοια ε, ε, ε, ιδιωτική εκπαίδευση. Πρέπει να βρεθεί μια νέα φόρμουλα, ένα νέος τύπος για να εφαρμοστεί στη σχολή της Χάλκης για το δημοκρατικό άνοιγμα, αληθεύει και η κυρία Φλότρο το είπε, δεν υπάρχει συνένεση προς το παρόν για να γίνει συνταγματική μεταρρύθμιση. Προσπαθεί η κυβέρνηση να έχει διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου αλλά ε, στο μεταξύ θα εγκρίνει ε, μεταρρυθμίσεις ε, για την διδασκαλία και για τις εκπομπές, ό,τι δεν χρειάζεται συνταγματική μεταρρύθμιση και τώρα δεν έχω άλλο χρόνο. Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση του κ. Χατζη Γεωργίου, γιατί σας έκανε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί χάλκι λέτε. όχι, λέει η Πρόεδρος, για την Κύπρο σας ρώτησε κάτι. The question η ερώτηση, κύριε Πρέσβη, για το 301, αν συμφωνείτε ότι πρέπει να φύγει και για την δίκη ενάντια στο κυβερνών κόμμα, πού βρίσκεται, διότι θυμούμε καλά ότι δεν έκλεισε. Επευλήθη ένα πρόστιμο, αν είναι δυνατόν, ενάντια στο κυβερνών κόμμα, αλλά παρέμεινε η δίκη. Θέλω να ξέρω πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Ambassador. Ε, κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Για το 301, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πολλές χώρες που διαθέτουν παρόμοιους νόμους και εμείς ακολουθήσαμε τα πρότυπα άλλων χωρών. Δεν νομίζω δηλαδή ότι απαιτείται η πραγματική πλήρης κατάργηση του 301. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση κατά του κυβερνώντο κόμματο, η δίκη αυτή ολοκληρώθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο και δεν, αναμένονται, δεν αναμένεται να αναλυθεί άλλη δράση. Η πρόεδρο. ναι, προφανώς ορισμένε άλλε χώρε έχουν παρόμοια άρθρα στους ποινικού κωδικέ του, αλλά εμείς εδώ στην υποεπιτροπή μας είμαστε απολύτω αντίθετοι, είτε πρόκειται για την Κίνα, τη Ρωσία, την Τουρκία. Θα ήθελα... Α, η κυρία Φλότ λέει η Γαλλία. Κύριε Φιλόρη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, μπορείτε να πείτε με λίγα λόγια πώς βλέπει η Επιτροπή την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Τουρκία. Και θα το, η δική σας παρέμβαση θα είναι και η τελευταία. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εγώ διαπιστώνω καταρχήν ότι πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στην έκθεση της Κομισιόν. Και λέω, ορίστε μια έμεση από τις τιμής ε, στις εργασίες ε, των ε, συναδέλφων μου. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία λέμε στην εκθεσή μας που δημοσιεύτηκε στις 14 Οκτωβρίου αλλά θέλω να καλέσω τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συνεδρίαση να ε, το έχουν καθαρά στο κεφάλι τους από πού ξεκινήσαμε στην Τουρκία. Δηλαδή είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα που ανταποκρίνονται στα αιτήματα τα οποία έχει ε, υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Συμφωνία Συνεργασίας και ορισμένες από τις εξελίξεις που μεσολάβησαν αποτελούν πραγματικά ένα χάσμα εναντί του παρελθόντος, ένα σπάσιμο πλήρες με το παρελθόν. Δηλαδή τα δικαιώματα, τα πολιτιστικά δικαιώματα, το ότι αναγνωρίζονται άλλες γλώσσες πλην της τουρκικής και μάλιστα 24 ώρες το 24ωρο ε, ένα δημόσιο κανάλι είχε εκπομπές στα κουρδικά. Επίσης είδαμε και ένα νόμο για τα οπτικακουστικά που καταργεί οποιοδήποτε περιορισμό στην ραδιοφωνική τηλεοπτική αναμετάδοση άλλων γλωσσών που να μην είναι τουρκική. Έτσι λοιπόν υπάρχει απόλυτη ελευθερία εκπομπή σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς υπότιτλους, χωρίς μεταφράσεις κλπ. Και ο... Για όποιους παρακολούθησαν ε, τα τελευταία χρόνια τα διαμηθέντα στην Τουρκία, πραγματικά πρόκειται για κάτι το φοβερό ως εξέλιξη. Τώρα οι άλλοι ομιλητές αναφέρθηκαν σε προβλήματα. Εμείς ε, στην Κομισιόν δεν διαφωνούμε στην ύπαρξη αυτών των προβλημάτων. Εμείς ε, όλα αυτά τα προβλήματα τα συζητάμε, έχουμε διάλογο με τις τουρκικές αρχές, ούτως ώστε να έχουμε και σημαντικές βελτιώσεις ήδη φέτος, ούτως ώστε του χρόνου να έχουμε ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα από ό,τι τα φετινά. Σας ευχαριστώ. Είμαι πεπισμένη ότι η ιστορία ε, της προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προϊούσα και την κυρία ε, ε, Φλότχοτ, κυρία Μενόρτον, θα τις προσκαλούμε πολύ συχνά στην υποεπιτροπή μας για να στοιχειοδετούν στις συζητήσεις μας, για να μας ενημερώνουν. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα συνεχίσουμε με μια συνεδρίαση και ε, των θύρων. Θα γίνει ε, ε, ενημέρωση με διαβαθμισμένες πληροφορίες για τις διαβουλεύσεις που έχει κάνει η Σουηδική Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να αποχωρήσουν όλοι πέρα από τα μέλη και το προσωπικό της Επιτροπής.